So. good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε στην συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σα σχίσουμε γιατί είναι τη και τέταρτο. Έχουμε καθιστήσει ένα τέταρτο. Πάνω στο σημείο 1, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Να ανακοινώσω ότι στο σημείο 6 τη ημερήσια διατάξεω για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το συζητήσουμε πριν το σημείο 5 για τη Συρία. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, η τροποποιηθήσα ημερήσια διάταξη θεωρείται συγκεκριμένη. Πάμε τώρα στο σημείο 2 ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν υπήρχαν κάποιε όταν συνετάχθη το κείμενο αυτό, ούτε από την πλευρά σα. Έχετε κάτι να πείτε. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των προηγουμένων. Είχαμε μία 13 Σεπτεμβρίου 2017. Έχετε σχόλια. Δεν έχετε. Πάμε στο σημείο 4, ενημέρωση όσον αφορά την αποστολή μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έλαβε χώρα 30 και 31 Οκτωβρίου του 2017 και αποστολή στη Ουάσιγκτον και στο Νόρφοκ στις 31 ε, Οκτωβρίου μέχρι 3 Νοεμβρίου. Η αποστολή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διεξήχθη όπως κάθε χρόνο μαζί με την Υποεπιτροπή Ντρουά, ενώ επίσκεψη στη Ουάσιγκτον, DC και στο Νόρφοκ πραγματοποιήθηκε από κοινού με τη ΣΕΝΤΕ. Τα βασικά θέματα τη επισκέψη στη Νέα Υόρκη ήταν η ειρήνη, η ασφάλεια, η πρόληψη συγκρούσεων, ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστευση και αλλαγή του κλίματο. Είχαμε παραγωγικέ συναντήσει με του ομολόγου μα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα, του κ. Αντώνιο Γκουτιέρε, του νέου Προέδρου τη Γενική Συνελεύσεω Μύρο Λάιτσακ, του Ενωπηρετού Γραμματέα για Πολιτικά Ζητήματα και του, της Διευθύνσεως για Ειρηνευτικές Αποστολές του ΟΗΕ και το πρόγραμμα του του ΟΗΕ να αναφέρω μερικέ πτυχέ. Είπαμε ότι υποστηρίζουμε τι μεταρρυθμίσει που πραγματοποιεί και ο Αντώνιο Κουτέρου, που δίνει μια νέα όθηση για ισχυρότερα Ηνωμένα Έθνη. επαναλάβαμε το βασικό ρόλο του ΟΗΕ να προωθεί πολυμερή προσέγγιση στα προβλήματα και προστασία των διεθνών κανόνων και αξιών. Απευθύναμε πρόσκληση στον νέο πρόεδρο τη Γενική Συνελεύσεω, τον κύριο Μιροσλάβ Λάιτσα, και είπαμε να έρθει σε μια συνεδριά τη ΑΦΕΤ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτου, του 2018. Οι επισκέψει στον Washington και τον Όρφολκ τη Βιρτζίνια ήταν καλποφόρε. Στον Όρφολκ επισκεφθήκαμε ε, το, την ε, συμμαχική δίκηση του ΝΑΤΟ και το τμήμα μεταρρυθμίσεων και συζητήσαμε τα θέματα κυβερνασφαλείας, υβριδικών κινδύνων και διάφορα τα θέματα. Επισκεφθήκαμε επίσης και τον αύσταθμο του Αμερικανικού Ναυτικού στο Νόρφολκ της Βιτζίνια. Στη Ουάσιγκτον, η αντιπροσωπεία μα συναντήθηκε με του συναδέλφου μα στο Κογκρέσο, όπου συζητήσει εστιαστήκαν ε, φυσικά στο Ιράν μετά την πρόσφατη απόσυρση τη εγκρίσεω ε, τη συμφωνία με το Ιράν και τα πιο ευρεία θέματα που αφορούσαν ε, τη σχέση Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Επίση, είχαμε συναντήσει το Πεντάγωνο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλεία, το Υπουργείο Εξωτερικών και είχαμε συζητήσει που ήταν σημαντικέ με διάφορε ομάδε προβληματισμού για τη διατλαντική ασφάλεια και τα Δυτικά Βαλκάνια και τη συνεργασία για τη διατλαντική ασφάλεια. Αυτά είχα να πω όσον αφορά τι επισκέψει Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον. Να δώσω σε κάποιου από του συμμετέχοντε σε αυτέ τι αποστολέ το λόγο και θα δώσω στον κύριο Παντζέρη το λόγο που είναι ε, ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής ε, Ντρουά. Έχετε το λόγο κύριε Παντζέρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας πράγματι, πράγματι. Τουλάχιστον όσον αφορά την επίσκεψη που ενδιαφέρεται την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχαμε συναντήσεις ε, σημαντικότατες, άκρως ενδιαφέρουσες και ήταν ε, πολύ καλή συνεργασία με τους ομολόγους μας και εμβαθύναμε σε διάφορα θέματα από μετανάστευση μέχρι θέματα, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητήσαμε. Όπως υπογραμμίσατε κι εσείς, ε, πολλές από τις ε, συναντήσεις επικεντρώθηκαν πάνω απ' όλα στο θέμα της μεταρρυθμίσεως του ΟΗΕ και πιο συγκεκριμένα στην αναδιοργάνωση στην εσωτερική περισσότερο που ήταν από τα σημαντικότερα στοιχεία δηλαδή λειτουργία του όλου μηχανισμού, ούτω ώστε να είναι πιο εκτεταμένες και αναγνωρίσιμες οι πολιτικές που εφαρμόζονται για το ξεπέρασμα της κρίσης εξοπιστίας ε, από το οποίο υποφέρει ο ΙΕΣ σε διεθνές επίπεδο. Είχαμε επίσης ε, σημαντική συνάντηση με την υπηρεσία του, του Επιτρόπου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και είναι χρήσιμο να σταθούμε επ' αυτού για να δώσουμε και κάποιες ενδείξεις να τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα. Ουσιαστικά στις συζητήσεις μας διεφάνει το εξή. Οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους λειτουργεί ο ΙΕ είναι η ανάπτυξη, οι ειρηνευτικές πολιτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, ε, εμείς ρωτήσαμε πότε θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός για τον τρίτο πυλώνα και η απάντηση που ήταν 3% ουσιαστικά για τη χρηματοδότηση. Δηλαδή θα είναι πολύ μικρή, μικρός πυλώνας σε σχέση με τις δραστηριότητε που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ΙΕΣ σε αυτό το τομέα. Πιστεύω από την πλευρά μας και από την πλευρά τους υπάρχει επίγνωση ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις προς τα εκεί, ε, συμφωνήσαμε μαζί τους ε, ή δυνατόν ετησίως να καθορίζεται ένα πρωτόκολλο μεταξύ της Υποπιτροπής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, το, και της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΕ όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις προοπτικές που υπάρχουν. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα του πρωτόκολλου του ετησίου μπορεί να γίνει ένα στοιχείο σημαντικότατο, ένα εργαλείο που μπορεί ε, να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για ένα θεματολόγιο μελλοντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε από ευρωπαϊκή άποψη να πούμε ότι εκεί συμβάλαμε. Δηλαδή γενικά πιστεύω ότι υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ ΑΦΕΤ και ΤΡΟΑ Η επίσκεψη θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη τελικά, θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για τις εργασίες μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στους ομιλητές των ομάδων. Μάικλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Α, μια στιγμή. Πρώτα Νέα Υόρκη και μετά Ουάσιγκτον. Εντάξει, καλύτερα μάλλον. Ε, ζητώ συγγνώμη, Μιχέλ. Bitte, Eugen Freund. Eugen Freund, να πει πρώτα για την Νέα Υόρκη και μετά στην Ουάσιγκτον. Ε, πάρα πολύ σύντομα στα αγγλικά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συνάντηση που είχαμε εκεί. Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερος, οφείλω να πω, από τις συζητήσεις που είχαμε με τον Τζέφρι Φέλτμαν, αναπληρωτή ε, υπουργών πολιτικών υποθέσεων. Ε, έθιξε σχεδόν όλα τα θέματα που μας απασχολούν και μας από την Ουκρανία, Συρία μέχρι τη Λιβύη Εξεπλάγει, ε, ακούγοντας αυτά που είπε, δεν τον παραθέτω, συνοψίζω, είναι πιο αισιόδοξο από εμάς για τη Λιβύη σε ό,τι αφορά την κατάσταση εκεί. Για τα Βαλκάνια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή αυτή, όπως και εμείς άλλωστε απομένουν πολλά να γίνουν και στην Ουκρανία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις και την πρόταση της Ρωσίας να επιτραπούν στρατεύματα εκεί ειρηνευτικά. Αλλά δεν έχει καταλήξει αυτό το θέμα, αν θα γίνει όχι. Για την Ιεμένη, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί και μας βρήκα ενδιαφέρον αυτό που είπε, ότι ενδιαφέρεται η Σαουδική Αραβία να τελειώσει εκεί ο πόλεμος, να τερματιστεί. Εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό, αλλά εκείνος μάλλον είναι πιο ενημέρος από μας. Αυτά σε γενικές γραμμές συνοψίζουν τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης, ιδιαίτερα και με το Γενικό Γραμματέα. Το είπατε και εσείς, Πρόεδρε θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση το σημαντικότερο παράγοντα σε αυτόν τον κατακαιρματισμένο κόσμο που ζούμε. Και παράγοντα σταθερότητας εννοεί. Και πραγματικά αυτό μας παρηγορεί να τα ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Άγγιν Φρόντ. Ο Γιώ Λάινεν επίσης για τη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Φρόιντ. σε μια συνεδρίαση ε, στη Νέα Υόρκη διαπιστώσαμε πόσο σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΟΗΕ. Ιδιαίτερα τώρα που επικρατεί νέα βεβαιότητα με την νέα Αμερικανική κυβέρνηση και ε, με διάφορες περικοπές ή ε, απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από διάφορα προγράμματα. Χρειάζεται βοήθεια ο ΙΕ και είναι σημαντικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά ένα πυλώνα τη υποστήριξη αυτή. Επίσης διαπιστώσαμε κατά τις συνομιλίε μας ότι η Κίνα και στα Ηνωμένα Έθνη ανεβαίνει, οργανώνεται, ισχυροποιείται όλο και περισσότερο στις συνευτικέ αποστολές αλλά και στα οικονομικά. Και βεβαίω είναι ευπρόσδεκτο κάτι τέτοιο. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν χρειάζονται μόνο υποστήριξη, χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις. Συγκλονίστηκα από ένα γεύμα που είχαμε με τρεις αρμοδίους για τις μεταρρυθμίσεις και η λέξη ε, δυσπιστία και καχυποψία ε, κυριαρχεί παντού στον ΟΗΕ. Ε, οι πάντες υποπτεύονται τους πάντες. Οι πάνω τους κάτω, οι κάτω τους πάνω, δεξιά τους αριστερά και πάει λέγοντας. Έχει εσωτερικά προβλήματα ο ΟΗΕ που θέλει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει ο Γενικός Γραμματέας με τις μεταρρυθμιστικές του προτάσεις δεν μπορούμε παρά να το ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία. Μας είπε επίση ότι η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να με ακολουθήσει. Ξέρετε ότι στα Ηνωμένα Έθνη έχουμε διάφορα μπλοκ τα οποία είναι το ένα απέναντι στο άλλο ε, ανυποχώρητα και ανένδοτα και ασυμφιλίοντα. Ελπίζουμε να τα καταλάβουν τα κράτη-μέλη αυτά τα μηνύματα, γιατί έτσι δεν αντέχει ο ΕΕ μέσα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία θα ε, υποχωρήσει στη δυνατότητα που θα έχει να λύνει συγκρούσεις και να ασχολείται και με νέα προγράμματα. Για τα νέα προγράμματα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Άχιμ Στάινερ, διευθυντής του προγράμματος για την ανάπτυξη, είναι δυναμικός. Το ξέρω και από την ε, παλιά θέση του στα προγράμματα UNEP ε, για το περιβάλλον. Και ξέρει πολύ καλά ε, με μικρούς, λίγους πόρους να κάνει αναπτυξιακή πολιτική που να πιάνει τόπο και στην Αφρική και άλλο. Και ένα στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο ΙΕ δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, για να μην πω ότι όλο και λιγότερα μπορεί να κάνει. Και περισσότερο θα πρέπει να ενέχονται εδώ περιφερειακοί ε, ε παράγοντες. Βλέπε Σαχέλ, ε, η Αφρική νοτίος ε, Σαχέλ Αφρικανική Ένωση και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πιο κοντινοί περιφερειακοί παράγοντες και μόνο έτσι μάλλον θα αντιμετωπίσετε. Το 2018 είναι το έτος της Ευρώπης στα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε πέντε κράτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γενικό Γραμματέα πρωτοφανή πράγματα αυτά. Το 2018 λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτή η χρονιά για τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια για τη Νέα Υόρκη. Ο τους παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τη σύντομη πληροφόρηση από τους συναδέλφους. Νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να παρακολουθούμε το τι γίνεται στον ΟΗΕ. Να... Εγώ δεν μπόρεσα να πάω με την αντιπροσωπεία, όμως ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες επερωτήσεις για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τις απαντήσουμε στη ορού της συζήτησης. Μιλήσατε για την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είμαστε και δεν μπορούμε από κοινού να δράσουμε, ε, θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω ε, ποια ήταν η δουλειά και πώς ε, μπορούμε να έχουμε πιο καλή δημοκρατική υπόσταση μέσα στα κρατημέλη, μέσα στα κοινοβούλια, στην κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και ακριβώς αυτή την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος να την προωθήσουμε. Και το δεύτερο ερώτημά μου, ε, το θέμα των προσφύγων αυτό το ζήτημα ε, και ειδικά ο, ο ρόλος που έπαιξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πόσο συζητήθηκε και πόσο συζητείται στον ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για τη Νέα Υόρκη. Να κλείσουμε λοιπόν. Δυστυχώς δεν είναι... Ο Άνρι Κόμπατζετ δεν είναι εδώ. Είναι ο εισηγητής μας και στην τελευταία έκθεση μαζί με τους Σκιώδης είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών. Το δεύτερο θέμα για την μεταναστευτική πολιτική το συζητήσαμε, παίζει ένα κεντρικό ρόλο. Ε, περίεργο που δεν υπήρξε στη συζήτηση με τον Άχεν στην οποία, η οποία εξελιχθήκε με τον Τζον Λάινεν για, την, για τον εκδημοκρατισμό του ΟΗΕ. Θέλεις να πεις κάτι? Die UNO ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Ε, τι κατατρέχει η εσωστρέφεια ε, τώρα αυτή ε, τη οργάνωση, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ε, ομφαλοσκοπή είναι μια μεταρρύθμιση προς το εσωτερικό, ενώ αυτό που λέει ο Χέλμουτ ε, Σόλτς είναι να δούμε αν υπάρχει μια νέα δυναμική με κινήσεις ε, έξωθεν. Στη Νέα Υόρκη είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι αυτό είναι δύσκολη υπόθεση πραγματικά η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Αλλά η κοινωνία των πολιτών, ε, τα κοινοβούλια και παγκόσμια κοινή γνώμη θα πρέπει να προσέχει περισσότερο τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αυτόν έχουμε, όσο προβληματικός και να είναι και δύσκολος, άλλο ο ΙΕ δεν έχουμε. Και δεν μπορούμε να έχουμε κανένα υποκατάστατο ερζάτσι ή να γεννήσουμε τίποτα καινούριο. Αυτό τον οργανισμό έχουμε. Και εμείς ε, ως Επιτροπή Εξωτερικών και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ντρουά και άλλοι, ε, και άλλες επιτροπές ασχολούμαστε. Είπε και ο Άχιμ Στάινερ ότι Έχουμε τα 75 χρόνια ε, σε τέσσερα χρόνια την επέτειο αυτή και ο Αντώνη Γκουτέρες ε, πραγματικά θα κρυθεί, θα κερδίσει ή θα χάσει από αυτό το πακέτο των μεταρρυθμίσεων. Το πρώτο, αν πετύχει Χιάλμουτ Σόλτ αυτό μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερο που να ε, φωτίζει, να ασχολείται με άλλες πτυχές. Μα είπα και εγώ στην αρχή, λέει ο Πρόεδρος, ότι σχεδιάζουμε ή τουλάχιστον θα προτείνουμε να έρθει ο πρόεδρος της 72ης Γενικής Συνέλευσης, ο Λάιτσεκ, ε, στην αρχή του 18 για να το συζητήσουμε. Και τονίζω αυτό που είπε ο Γιώ Λάινεν, ως Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχουμε μια σπάνια ευκαιρία, διότι είναι Ευρωπαίος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του χρόνου από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα 5 θα είναι ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τόσο πολύ Ευρώπη στην ηγεσία του ΟΗΕ είναι σπάνιο και μάλιστα πρωτοφανές. Και ο Αντώνη Γκουτέρες θέλει να είμαστε η σημαντικότερη σύμμαχοι του για να προωθήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Γιν Φρόιντ, ξαναζήτησε το λόγο. Μια πρόταση μόνο για τα θέματα του προσφυγικού ε, που μίλησε και ο κύριος Σόλτς για αυτό, ρώτησε. Φυσικά μας απασχολούσαν σχεδόν σε όλες ε, τις συναντήσεις μας ε, και πιο εύγλωτο είναι αυτό που μας είπε ο νυν πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ότι εκεί θα κρυθούμε, αν θα καταφέρουμε το πρόβλημα αυτό να το... Δεν είπε να το λύσουμε, νομίζω είπε να ε, το αντιμετωπίσουμε, να το ελέγξουμε, που είναι σημαντική διαφορά, όχι να το λύσουμε. Ε, να το πω τώρα. Γίνεται μια προσπάθεια να ε, ελέγξουμε ένα πρόβλημα το οποίο μας έχει όλους συγκλονίσει. Και μας αφορά πάρα πολύ. Και μας είπε ότι η αποτυχία δεν είναι επιλογή. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να αποτύχουμε, δεν το διανοείται κανείς αυτό. Failure is not an option. Αυτά. Thank you. We now come to the Washington. Ευχαριστώ. Πάμε στη Washington. Ο Μάιχελ Γκάλλορ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ για αυτή την ε, επίσκεψη ότι δεν συναντήσαμε τον ε, αρχηγό, ας πούμε, τον ύπατο υπάλληλο εκεί. Ήταν όμως επικοδομητική η συνάντηση γιατί συζητήσαμε τα περισσότερα θέματα και είδαμε ότι είχαμε κοινά στοιχεία. Ας πούμε στο θέμα του Ιράν εμείς είπαμε ότι έναντι του State Department του Πενταγώνου των δύο ε, σωμάτων του Κοινοβουλίου είπαμε ότι περιμένουμε οι Ηνωμένε Πολιτείες να τηρήσουν τη συμφωνία για τα ατομικά όπλα. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία ε, έχουν να κάνουν πούμε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιρροή στην περιφέρεια αυτή, όλα αυτά που σχετίζονται. Λοιπόν, θα πρέπει ε, να τα συζητήσουμε και αποκοινούμε κοινού τις ΗΠΑ να δράσουμε εναντί του Ιράν ο Άνοκ επίσης ε, ήταν ένας από τους ρεπουμπλικανούς ε, που συναντήσαμε. Δεν ήταν 100% κατά, κατά της συμφωνίας δηλαδή. <clears throat> Δεν θεωρεί ότι είναι μια κακή συμφωνία, όμως είπε συγκεκριμένα ότι είναι καλύτερα να έχουμε αυτή τη ε, συμφωνία για να μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να μπορούμε να τους ελέγχουμε. Επίσης, ήταν θετικό το νέο ότι όταν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο άμυνας, ε, κανείς δεν θα εναντιωθεί, θα μας υποστηρίξουν. Από την, κατά την άποψή μου λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Είμαστε λοιπόν στο δρόμο μιας ενίσχυσης της θέσεις της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ, ε, να μπορούμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική συνεργασία. Για τη Βόρεια Κορέα επίσης ε, και πάλι τέθηκε το θέμα με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Φυσικά η διπλωματική λύση είναι η πρώτη επιλογή. Επίσης, ε, υπόθηκε ότι ε, το γεγονός ότι ο πρόεδρος ε, χρησιμοποίησε σκληρά λόγια είχε να κάνει με, το, με τη σχέση του με τον Κιμ Γιονκούν. Είναι ο τρόπος που εξελίσσεται η διπλωματική συζήτηση. Στο Πεντάγωνο βέβαια δεν έβγαλε και μεγάλο συμπέρασμα όταν μας είπαν ότι είμαστε τελευταίοι που θέλουμε τον πόλεμο. Όταν το λέει αυτό ένα Υπουργείο Άμυνας δεν ξέρω κατά πόσο είναι επικοδομητικό, αλλά σίγουρα ε, η διπλωματία είναι πρώτη. Αυτά είχα να πω για τα τρία βασικά θέματα που συζητήσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κουρτ Φλέκενστεν. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ε, επαναλάβω αυτά που είπε ο Μίχαλ Γκάλερ. Συμφωνώ ότι πραγματικά ε, επεκταθήκαμε σε πολλά θέματα ειδικά στο State Department, για την περιοχή του Κόλφου, την Τουρκία, την ε, πάταξη της ε, τρομοκρατίας. Ε, νομίζω ότι υπήρξε καλή ανταλλαγή απόψη, απόψεων και ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι οι φίλοι μας οι Αμερικανοί στο State Department. Για το Ιράν επίσης, νομίζω ότι οι Αμερικανοί έχουν μια πολύ εντυπωσιακή αποφασιστικότητα από το ECR μέχρι τον ΚΟΕ όλοι. Ε, είπαμε, μιλήσαμε με τον ίδιο τρόπο ε, για το Ιράν. Κανείς ε, δεν διαψεύδει ότι υπάρχει μια σειρά προβλημάτων με το Ιράν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όμως αυτή η συμφωνία, η λεγόμενη Run Deal, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστραφεί. Δεν πρέπει να τη βλάψουμε. Επίσης, ε, υπήρξαν συγκεκριμένες τρεις απαντήσεις για την προσέγγιση που έχουν οι Αμερικανοί. Ε, δεν το θέλει ο Πρόεδρος. Ε, δεν είναι ξεκάθαρο αν τελικά θα τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά γενικά εμείς ε, το δείξαμε πολύ ξεκάθαρα ε, και εξετάσαμε και κατά πόσο μέσα από κάποια συμπληρωματικά πρωτόκολλα θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις. Ε, επίσης, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο το Ιράν έχει πραγματικά κατά 100% εκπληρώσει τα όσα εγγράφονται στη συμφωνία. Κάτι άλλο που και εγώ θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την πολύ καλή προετοιμασία για τη δουλειά, ειδικά επειδή υπήρχαν πάρα πολλά που έπρεπε να κάνουν και όλα πήγαν πολύ καλά. Τους ευχαριστώ. Επίσης, να πω ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι καλό. Έχουμε επαφές και καλές επαφές, όμως πρέπει να δούμε, να βρούμε έναν τρόπο καλύτερα να συμφωνούμε και να συντονιζόμαστε. Ήταν πολύ καλό το ταξίδι μας. Ε, θα ήταν ακόμα καλύτερο ε, αν υπήρχε καλύτερος συντονισμός των ταξιδιωτών και εγώ δεν είχα ε, ε, κάποιο πρόβλημα, αλλά στο Προεδρείο ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο ε, Φλέκενστάιν. Μετά και στο επόμενο Προεδρείο θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θέλουν να πούν κάτι. Αν όχι, να σας πω ότι εχθές είχα την ευκαιρία με την κυρία Μοργκερίνη να τηλεφωνηθώ και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την Ουάσιγκτον. Και αυτή θα πάει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον και θα συζητήσει και το Ιράν με τον Μάικ Πρέντς, τον αντιπρόεδρο. Και της είπα ξεκάθαρα ότι η δική μου εντύπωση ήταν πως ε, οι Αμερικανοί ήταν ιδιαίτερα θετικοί, έδειξαν κατανόηση και με εντυπωσίασε ε, πόσο μεγάλη αλληλεγγύη υπάρχει για αυτό το θέμα από το ECR μέχρι και το, και το άλλο άκρο ε, του φάσματος για όλα τα κόμματα. Επίσης ε, για τον τομέα αυτό κάθε φορά που μπορούμε θα πρέπει να τονίζουμε πως πρέπει να τηρηθεί το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, συμφωνία με τον Ιράν. Επίσης να ευχαριστήσω και εγώ για την προετοιμασία. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο, ο Γκεν Δεν θέλω να αφήσω να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, επειδή δεν το είπε κανεί. Και το λέω λοιπόν ρητά αυτή τη στιγμή ότι και εμεί είμαστε ικανοποιημένοι με την προετοιμασία, την διεξαγωγή και την προεδρία. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ε, αποστολή. Σας ευχαριστώ για τους ε, ευγενικούς σας επένους και προς την γραμματεία βεβαίως και τη γραμματεία ΣΕΝΤΕ και Ντρουά παρακαλώ να τα διαβεβάσετε αυτά ε, και μιλώ εξ ονόματος όλων των παρόντων και των συμμετεχόντων. Αν δεν έχουμε τίποτα άλλο να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα το που έχουμε προτάξει και είναι το 6, πρώην 6 νυν 5 και μάλιστα επιγράφεται το εξής. Θα συζητήσουμε λοιπόν το σχέδιο νομοθέτηση τη ΑΦΕΤ όσον αφορά την προετοιμασία του υπολογισμών για τη θέση του Κοινοβουλίου για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020. Βεβαίω είναι σημαντικό το τομέα όπου η Επιτροπή μα θα περιγράψει τι προτεραιότητέ τη για τη χρηματοδότηση τη βοηθεία και δράσεων για την υποστήριξη εξωτερικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, συμπεριλαμβανομένε τη διευρύσεω και πολιτική γειτονία. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Παντζέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με αυτό το σχέδιο γνωμοδοτήσεως η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να δώσει κάποιες ενδείξεις όσον αφορά τον προπολογισμό για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως και μετά το 2020 θα υπάρξουν πολλά προβλήματα και προκλήσεις. Θα πρέπει μετά το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ενσαρκώσει ε, τη δήλωση που έχουμε κάνει, δηλαδή να είμαστε μεγάλοι για τα μεγάλα ζητήματα και ε, μικροί για τα μικρά θέματα. Λοιπόν, στη χρηματοδότηση τόνισα τρία βασικά σημεία. Πρέπει να αυξηθεί ουσιαστικά η χρηματοδότηση για την εξωτερική δράση στόχος η εξωτερική πολιτική και η εξωτερική πολιτική να είναι θεμελιώδης λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην αναπτυξιακή βοήθεια, προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προώθηση του κράτους δικαίου, δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές κατά της ασφάλειας, την αποφυγή ενόπλων συγκρούσεων, την τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές, κακή ε, διοίκηση, ε, ανταλλαγή του κλίματος, και όλα τα προβλήματα που αναδύονται. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Και έτσι μπορούμε να κινητοποιούμε πόρους για ανταπόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Χωρίς όμως να υπονομεύουμε την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων με τη μείωση άλλων χρηματοδοτήσεων. Τέλος, ε, όσον αφορά τα ταμεία που δημιουργήσαμε όπως αυτό για την Αφρική και τη συμφωνία με την Τουρκία, θα πρέπει αυτά τα ταμεία να μην χρηματοδοτούνται μέσω της μειώσεως πόρων που προορίζονται σε άλλες δράσεις. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος ο πλευράς των φορέων του προπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου. Για λόγους χώρου δεν μπορέσαμε να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Το κείμενο θα λάβω υπόψη τροπολογίες, καλώ τις ομάδες μέχρι 23 Νοεμβρίου να υποβάλουν τροπολογίες. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Παντζέρη. Πάμε τώρα στα σχόλια των σκιωδών εισηγητών. Κρίστιαν Πρέντα μου τηλεφώνησε το πρωί και μου είπε να διαβάσω τη δήλωσή του. Με τα χαράς. Λέει λοιπόν, καταρχάς εκφράζω τη λύπη μου που δεν μπορώ να είμαι παρόν στην πρώτη συζήτηση το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι επίκαιρο θέμα για την Επιτροπή μας, θα πρέπει να σε ακουστεί η φωνή μας στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Το παρόν πολιτισμικό συνικό πλαίσιο έδειξε ότι έχει όρια τα τελευταία χρόνια στον τομέα εξωτερικών υποθέσεων που επλήγει ιδιαίτερο από αυτή την έλλειψη. Υπό το φω των διαφόρων κρίσεων που αντιμετωπίζουμε, ότι δεν διατίθενται αρκετοί πόροι. Αυτό είναι φανερό για, ε, για το πολιτιστικο για το πολιτισμικό πλαίσιο 2014-2020 και οι μηχανισμοί ευελιξία παραδόξω δεν ήταν αρκετά ευέλικτοι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά μηνύματα που πρέπει να στείλουμε μέσω τη γνωμοδοτήσεω και χαίρομαι ιδιαίτερω που βλέπω ότι η μα, ο κ. Αντώνιο Παντσέρη, έχει διάποψη. Δεν μπορούμε αξιόπιστα να διατηνόμεθα ότι προσπαθούμε να λύσουμε τις παρούσες κρίσεις στη γειτονιά μας και αλλού αν τις φιλοδοξείς πολιτικές δεν τις χρηματοδοτούμε επαρκώς. Ε, ο τομέα εξωτερικών υποθέσεων και η κοινή άμυνα γίνονται αντιληπτέ ότι έχουν μεγάλη δυνατότητα για προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία αν αντιμετωπιστούν σωστά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και όχι σε εθνικό. Μπορούμε να είμαστε πολύ πιο επιτυχεί και να εξασφαλίζουμε εξωτερική ασφάλεια για του πολίτε, προωθώντα την ειρήνη, αν συνδυάσουμε του πόρου μα ε, και έχουμε και καλύτερη συνεργασία μεταξύ μα. Δοθισών των συζητήσεων που κάνουμε τώρα για του προσανατολισμού του προπολισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, για να χρηματοδοτούνται οι μηχανισμοί που δίνουν προστιθέμενη αξία. Εδώ ζητούμε σημαντική αύξηση του κεφαλαίου 4, του τμήματο 4. Θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε για την σωστή ισορροπία μεταξύ προβλεψιμότητα χρηματοδοτήσεω και ευελιξία, όπω Είδαμε ότι τα τελευταία 7 χρόνια ε, σημειώθηκαν απρόβλεπτα γεγονότα που πρέπει να απαντηθούν. Η προσφυγική κρίση άσκησε πολλέ πιέσει στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, κυρίω όσον αφορά διάφορε πολιτικέ που επλήγησαν, διότι δεν είχαμε μια ένα απόθεμα για τη μετώπιση των κρίσεων. Τέλο, θα πρέπει γρήγορα να, υπογραμμίσουμε, να υπογραμμίσουμε, υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θα πρέπει να ακολουθήσουμε ε, σωστή πορεία. Οι υποτροπολογίε εστιάζονται επί ενισχύσεως τριών μηνυμάτων που θα πρέπει να στείλουμε. Ε, και θα έχουμε άριστη συνεργασία με τον εισηγητή. Θα στείλουμε σαφές μήνυμα την Επιτροπή μας για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Υπογραφή. Κρίστιαν Πρέντα. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Γκουε NGL. Κυρία Λόιζεν, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κάποιες ε, βασικές διαφωνίες, για να μην πω πολλές βασικές διαφωνίες, ως προς τον προσανατολισμό το γενικότερο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Εμείς τα βλέπουμε αυτά κυρίως, ε, να μην πω αποκλειστικά, στον πολιτικό τομέα, κατά πολέμηση της ένδυας, ανθρωπιστική βοήθεια, επίγουσα βοήθεια και ακόμα περισσότερα. Εμείς θέλουμε αμυγός πολιτική, εξωτερική πολιτική και διπλωματία. Και διαβλέπουμε τον εξή κίνδυνο τώρα εδώ. Με τα νέα προγράμματα, το πρόγραμμα για την αμυντική έρευνα και την υποστήριξη εξοπλιστικών ε, προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πολιτική ειρηνευτική ε, διάσταση. Κύριε Παντσέρη, εσείς μιλάτε για πολλά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτυξιακή πολιτική, κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, στη τελική ανάλυση, όταν λέτε για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, χρησιμοποιείτε έναν όρο, ε, ανανεωμένη, renewed. Τι σημαίνει αυτό. Εμείς λέμε νέο προσανατολισμό, όχι να ανανεώσουμε την πολιτική γειτονία. Ένα νέο προσανατολισμό θέλουμε και μας λείπει από την έκθεση αυτή αναφορά. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα όπως παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπανάπτυξη, ένοπλες σειράξεις που είναι συνέπεια της πολιτικής γειτονίας και εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον έτσι το θεωρούμε εμείς με τις αμυντικές και εξοπλιστικές δαπάνες που αποφασίζονται δεν θα σταθεροποιήσουμε τη γειτονία, το, αντί, το αντίθετο, θα έχουμε ε, περαιτέρω στρατιωτικοποίηση. Παρ' όλα αυτά, το σημείο 4 της νομοδότησης το υποστηρίζουμε ακόμα και αν στα ε, καταπιστευματικά ταμεία έχουμε πολύ μεγάλες αμφιβολίες ε, και γενικά τα απορρίπτουμε, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτών των ταμείων σε περίπτωση που περάσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λέζεν. και ο κύριο Καστάλντο από την ομάδα EFTD. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Παντσέρη, έξοχη δουλειά που έκανε στη σύνταξη του κειμένου. Εκτιμούμε τα μάλα τη σημασία ολιστικής προσεγγίσεω μακροπρόθεσμη, ούτω ώστε να στηριχθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως όταν προβλέπονται μηχανισμοί ευελιξία για την κινητοποίηση πόρων σε περιπτώσει απρόβλεπτες και κατεπίγουσες. Αυτή η ευελιξία, όπως έλεγε ο δεν θα πρέπει να είναι ει βάρο των στόχων των μακροπρόθεσμων που καθορίζονται τι πολιτικέ, τι ειδικέ και συγκεκριμένε. Πρέπει να αυξηθούν οι πόροι όσον αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτω ώστε η Ευρώπη να γίνει φορέας που να μπορεί να αντιμετωπίσει τι παγκόσμιες προκλήσει ε, κυρίω για την πολιτική γειτονία, τα αναγκαία μέσα, αύξηση για την αναπτυξιακή βοήθεια, τη διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σημείο 4 σημαντικό, να υπάρχει έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα καταπιστεύματα, τα trust funds και το Europe Facility for Refugees in Turkey. Είναι μια συμφωνία αυτή που ε, πάντα είμαστε εναντίον, δεν την εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει κατά την άποψή μα να τίθεται υπό τον έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου. Και το σημείο 5 είναι σημαντικό, υπό τη φω τη Ανατολική και νότια γειτονιά αντιμετωπίσουμε τα αίτια της, των προβλημάτων σταθερότητα, που τα προβλήματα οδηγούν και στα μεταστευτικά προβλήματα. Τέλο. όσον αφορά την προεντεξιακη βοηθεια βοήθεια, pre-accession, όσον αφορά την Τουρκία, που έχουμε μεγάλο προβληματισμό γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, βλέποντα και τι εξελίξει εντό τη Τουρκία, είμαστε υπέρ τη ενισχύσεω του πρωταξιακού μέσου. Θα πρέπει λοιπόν να ευνοήσουμε την πρωταξιακή βοήθεια προ τι χώρε όπω είναι το Μαυροβούνιο, που κάνουν σημαντικά βήματα πρόοδου, εφαρμόζοντα σωστά και ισορροπημένα όχι μόνο το κριτήριο του, του more for more, αλλά και του less for less. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Σίγουρα θα είναι πολύ καρποφόρος οι εργασίε που θα κάνουμε και θα οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Δύο ομιλητέ έχουμε ακόμα. Έναν από το ΕΛΚ και έναν από το EFTT. Ο Έντουαρτ Κούκαν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Ευπρόσδεκτο το σχέδιο γνωμοδοτήσεω του κυρίου Παντζέρη. Είναι ήδη πολύ καλό έγγραφο ως έχει και πολύ καλή βάση για παραγωγή του καλύτερου δυνατού εγγράφου που θα είναι αποτελεσματικό. Είναι σημαντικό να καθορίσουμε προτεραιότητες για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ευθύ εξ αρχή. Ευπρόσδεκτη λοιπόν η έκκληση για αύξηση των πόρων και για μεγαλύτερη ευελιξία και σχετικούς μηχανισμούς για εξωτερικά μέσα στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι σαφές ότι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και, τα, και την εξωτερική δράση θέλουμε να εφαρμόσουμε, θα πρέπει να πολεμήσουμε για αύξηση της χρηματοδοτήσεως για τα εξωτερικά αυτά μέσα. Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου. Συμφωνώ. Δεν θα πρέπει να ανακατατάξουμε τους πόρους για λόγους πολιτικούς. Καλύτερο θα ήταν να επικεντρωθούμε επί του αντιχτύπου που έχουν οι πόροι, να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων πολιτικών στόχων. Τα μέσα πρέπει να ταιριάζουν με τις τωρινέ και μελλοντικές προκλήσεις και σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά όλος ιδιαίτερος στη γειτονιά μας και στις χώρες ένταξης. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι πολιτικοί μας στόχοι συνάδουν με τα χρηματοπιστωτικά μέσα αυτό ισχύει ιδιαίτερως στους πολιτικά ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η γειτονία και η ένταξη. Κάτι που ήδη αναφέρθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Έντουαρντ Κούκαν. Και ο James Κάρβερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σε εκπλήσει που λέω ότι οι στόχοι εξωτερικής πολιτικής ε, με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Θέλετε να δώσετε περισσότερα χρήματα για στενότερη ένωση. Άρα για αυτούς σαν και εμένα στη χώρα μου που θέλουμε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και να πάμε για δεύτερο δημοψήφισμα μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Διότι εδώ γίνεται πιο στενή σχέση στην Ένωση. Λοιπόν, αν ήταν και να αλλάξει η άποψη η Βρετανία που φεύγει, θα ήταν δύσκολο αν θέλαμε να κάνουμε να αλλάξει η Βρετανία. Γιατί τώρα πάμε προς ε, Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Διότι αυτό δείχνει και αυτή η έκθεση. Και είναι και ελέφαντα στο δωμάτιο που δεν αναφέρουμε. Ε, δηλαδή, ότι θα φύγει η Βρετανία το 2020 που είναι ο τρίτος συνεισφορέας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα θα φύγουν τα 12% των πληρωμών για το προϋπολογισμό. Και αυτά προτείνεται είναι βραχυπρόθεσμες λύσεις. Πρέπει τελικά όμως τα λόγια να γίνουν χρήμα. Δεν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας που πληρώνει φορολογούμενοι από τα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση με άλλα λόγια. Αλλά να μην έχετε λιγότερες φιλοδοξίες, να μην έχετε απεικιοκρατικές ε, φιλοδοξίες και να μην θέλετε να επιβάλλετε τις απόψεις σας δικτατορικά στον υπόλοιπο κόσμο. you, Ευχαριστούμε τον James Carver. Έχουμε άλλον έναν ομιλήτη. Κύριε Σάφερτζερ, έχετε το λόγο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την αποτελεσματικότητα ε, της υποστήριξης της ανάπτυξης. Ε, βλέπω ότι σε πολλές χώρες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της παίζουν ένα ρόλο που δεν παίζουν άλλες χώρες. Δηλαδή αναλαμβάνει ενισχύσεις που δεν μπορούν να δώσουν άλλες χώρες. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ειδικά το Ταμείο Μακροπρόθεσμης Χρηματοδότησης που υποστηρίζει την, τις δραστηριότητες ανάπτυξης στην Αφρική ε, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντιθέτω, ε, θεωρώ ότι όσον αφορά τους μηχανισμούς ε, διεύρυνσης, αυτή τη στιγμή που και εμείς οι ίδιοι ακόμα δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε στο επίπεδο της Ευρώπης, κάνουμε, προτρέχουμε τέλο πάντων και θέλουμε καλύτερα θα ήταν να εξετάσουμε το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουμε ε, στην πολιτική της διεύρυνσης. Είναι δύο διαφορετικές πολιτικές λοιπόν. Ε, μιλάμε για αποτελεσματικότητα όσον αφορά στην ανάπτυξη και πώς η Ευρώπη θα μπορεί να συμπληρωματικά να δρά με την υποστήριξη των κρατών και από την άλλη έχουμε την πολιτική της διεύρυνσης η οποία αυτή τη στιγμή μου φαίνεται, πώς να το πω, πέραν της πραγματικότητας, πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ε, είναι, κάνουμε, προτρέχουμε και δεν ε, αντιστοιχεί αυτή η πολιτική στις πολιτικές που θα έπρεπε κανονικά να εκτελούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο σχόλιο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα στο ενδεικτικό ε, χρονοδιάγραμμα 12 ε, Νοεμβρίου στις 11 23 Νοεμβρίου στις 11 η, η πρωτοθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, τον ε, Γενάρη στις 22 θα έχουμε στην Βασική Επιτροπή την ψηφοφορία. Κύριε Παντζέρη θέλετε να πείτε κάτι, δεν σας είδα. Συντομότατος. Ευχαριστώ προφανώς όλους που παρενέβησαν. Θα συνεργαστούμε καρποφόρα λαμβάνοντας υπόψη τις υπενθυμιστής ε, προθεσμίες. Στο συνάδελφο Λόζινγκ να πω ότι ίσως τα λόγια στα Ιταλικά ίσως έχουν μερή έννοια. Όταν μιλάμε για ανανεώσιμη ε, ε, η λέξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί σαν κάτι διαδραστικό ή να εφαρμόζεται η ίδια πολιτική ή όπως θέλω να το πω εγώ ότι είναι κάτι ανανεώσιμο να αλλάξει κάτι επιρχαιωμένο δηλαδή το ανανεώσιμο πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση αν δεν λειτουργεί αυτή η λέξη ετοιμολογικά μπορούμε να βρούμε άλλη για να αποδώσουμε και το νόημα εκείνου που ήθελε να πει ο μιλητής στην παρέμβασή του. Okay, thank you. Any Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Όχι. Τώρα τελειώσαμε από σχόλια, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Στο σημείο 5, πρώην και νυν 6, παρακαλώ το προσκεκλημένο μας να έρθει στο Προεδρείο. Once again, welcome. You're familiar with the Okay. Okay, we now come to item number ε, Πάμε λοιπόν στο σημείο 5 και μεγάλη χαρά καλωσορίζω στην Επιτροπή μας τον κύριο Άντρου Τέιμπλερ από το Ινστιτούτο Ουάσιγκτον. Είστε ειδικό για τη Μέση Ανατολή και εργάζεστε επί σειρά ετών για στα θέματα της Συρίας. Την περασμένη εβδομάδα, όπως ακούσατε, πήγαμε στην Ουάσιγκτον ε, και στη Νέα Υόρκη. Ε, συζητήσαμε την κατάσταση στη Συρία, ιδιαίτερα με τον κύριο Γκουτέρες. Καταλαβαίνετε ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά και στενά τις πρόσφατες εξέλιξεις. Στις 22 Οκτωβρίου τερματίστηκε η κατάληψη της ΡΑΚΑ από τον ΤΑΕΣ, το Ισλαμικό κράτος, χάρη στις προσπάθειες διεθνούς συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό γιατί μειώνεται ο κίνδυνος και η απειλή. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος της Συμμαχίας ε, της Διεθνούς ε, συνεργάζεται με χώρες της περιοχής για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και γενικότερα ε, προγράμματα για, κατά της ρίζοσπαστικοποίησης. Είμαστε μάλιστα και ένας από τους βασικούς ηγέτες στη χρηματοδότηση. Υποστηρίζουμε το μέλλον της Συρίας στην περιοχή. 9,4 δις ευρώ έχουμε υποσχεθεί από το 2011 και σε αντίστοιχη διεθνή διάσκεψη που έγινε τον Οκτώβριο. Τώρα ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στη Ράκα και στην επαρχία συνολικά και πώς θα βοηθηθεί ο κόσμος μόνιμη ειρήνη βέβαια θα έρθει μόνο με τις συνομιλίες στη Γενέβη των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Τέιμπρερ, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για την πολιτική κατάσταση στη Συρία και ιδιαίτερα τις πολιτικές επιλογές τώρα που ανοίγονται για τη χώρα. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας δίνω μέσω στο λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, Πρόεδρε Μακάλιστερ. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που μου διαθέτετε σήμερα το χρόνο σας. Να ευχαριστήσω επίσης και την ε, αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με βοήθησαν για να έρθω εδώ σήμερα να σας μιλήσω για ένα επίκαιρο θέμα. Ένα θέμα που αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη γενικότερα. Έχουμε κοινό ε, ενδιαφέρον. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτει όταν μιλάμε για την Συρία ε, είναι σίγουρα ε, κατά πόσο αυτή, αυτό το ζήτημα επηρεάζει την πολιτική των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και αν σχετίζεται με αυτή. Θα ξεκινήσω με λίγα καλά νέα. Υπήρξε στρατιωτική ήττα του ISIS, του Ισλαμικού κράτους, ε, η οποία προχωρά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπαμε. Δυστυχώς βέβαια η πραγματική ήττα της οργάνωσης αυτής, δηλαδή το να φύγει τελείως ε, από το προσκήνιο, ε, δεν είναι και τόσο πιθανή, διότι τα βασικά ζητήματα που υπάρχουν στη Συρία ε, δεν έχουν επιληθεί. Δεν είναι ακριβώς έλλειψη δημοκρατίας, είναι έλλειψη συμμετοχής, απόλυτη έλλειψη κράτους δικαίου, λογοδοσίας και σε πολλούς τομείς σε πολλές ε, περιοχές της Συρίας, ε, σουνιτικές κυρίως, υπάρχουν ε, και μεγάλα δημογραφικά κύματα που πηγαίνουν πηγαίνουν προς τη Συρία και προς το Ιράκ. Ειδικά λοιπόν ο σεχταρινισμός ο σουνητικός έχει αυξηθεί. Υποστηρίζεται και από την κυβέρνηση του Ιράκ και από το καθεστώς του Ασάντ. Τα κακά νέα τώρα είναι, να μένω ότι χάνει έδαφος ο Άισις, αλλά το κενό που μένει πίσω το εκπληρώνουν οι Ρακινές στρατιωτικές ε, μονάδες και παραστρατιωτικές μονάδες, αυτές ε, που έχουν δημιουργηθεί για να, να μαχηθούν κατά του ISIS. Υπάρχει ε, μια εκτίμηση που ακούσαμε πριν από 15 μέρες. 80% των δυνάμεων που αυτή τη στιγμή μάχονται κατά του Ισλαμικού κράτους στην ε, Ανατολική ε, Συρία, που είναι μια κόκκινη βούλα στο χάρτη, είτε είναι χρηματοδοτούνται, είτε τις έχει οργανώσει το Ιράν. Αυτό δυστυχώς μας κάνει να ανησυχούμε. Τι είναι πίσω από αυτά. Ένα ερώτημα. Επίσης είναι και ανάγκη, διότι ε, το καθεστώς Ασάντ δεν μπορεί να ανταποκριθεί με ανθρώπινο δυναμικό, ε, διότι ε, έπρεπε εξ αρχής να διαθέσει πολύ ανθρώπινο δυναμικό για αυτή την κρίση και φυσικά με τον σεχταρισμό που υπάρχει δεν μπόρεσε να αναπληρωθεί. Ε, το Ιράν το υποστηρίζει επίσης η αεροπλοεία της Ρωσίας, ε, η οποία έχει βοηθήσει στην ανακατάληψη εδαφών. Βέβαια αυτά είναι μέσα από παρατηρήσεις, ε, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά βλέπουμε και αντιδράσεις στην Ανατολική Συρία που στην ουσία φαίνονται στον τοπικό πληθυσμό. Γιατί πηγαίνει ο τοπικός πληθυσμός ε, προς τις ε, ε, δυνάμεις του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού προς που υποστηρίζεται από τη Δύση και όχι, από τον, και όχι προς την πλευρά του Ασάντ. Αυτό μας επιβεβαιώνει ότι πραγματικά η υποστήριξη των κουρδικών δυνάμεων δεν είναι κάτι που θέλουν να δεχτούν οι ντόπιοι και επίσης ούτε και το καθεστώς του Ασάντ το προαραβικό περίπου ε, τελικά καθεστώς. Άρα φαίνεται πως ε, για να ξεφύγουν από τον ISIS πηγαίνουν πιο, πολύ προς τις δυτικά υποστηριζόμενες δυνάμεις. Τώρα ο πόλεμος ε, στην Συρία δεν έχει να κάνει μόνο με τον ISIS και στην Δυτική Συρία και στην, στις περιοχές του Ιράν όπου γίνονται οι εχθροπραξίες ε, έχουμε παρατηρήσει και έχουμε συζητήσει με τους διπλωματικούς εταίρους μας ότι η Τουρκία μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι του Συριακού πολέμου. Τους επόμενους μήνες λοιπόν θα περιμένουμε να επεκταθεί αυτή η προσπάθεια εν ώψη και μιας επίθεσης στρατιωτικής στην Άνοιξη για να, ε, μπορέσουμε, να, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ε, δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ειδικά αυτές που υποστηρίζονται από την Αλκάιντα. Τέλος, ε, υπάρχει η, συμφωνία στην νοτιοδυτική Συρία για την οποία, αποκλιμάκωση, η οποία φαίνεται ότι κρατάει και αυτό είναι καλό όμως ε, ε, τίθεται, τίθεται να αμφιβόλω η βιωσιμότητά της ε, λόγω των τοπικών ντόπιων δυνάμεων που δρούν και όσο περισσότερο μπαίνει το Ισραήλ σε αυτή την σύραξη. θα πρέπει να παρατηρήσατε ότι το καθεστώς της Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και η κυβέρνηση ανησυχούν ε, για την εξέλιξη του Συριακού πολέμου, ειδικά όσον αφορά στα δικά του σύνορα, γιατί υπάρχει μια τάση να ευνοείται η θέση του Ιράν. Ε, βέβαια, αυτό, αυτή η αποκλιμάκωση έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή. Συνολικά η ανθρωπιστική κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, πάνω από 500.000 άνθρωποι είναι αγνοούμενοι, 250.000 ε, έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, 4,8 ε, εκατομμύρια καταγεγραμμένοι πρόσφυγες ε, στις γειτονικέ χώρες, 1,5 εκατομμύριο εδώ στην Ευρώπη και άλλα 6,6 εκατομμύρια εκτοπισμένων εντό της Συρίας, ειδικά στις περιοχές όπου, όπου κυριαρχούν οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ε, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κρίση στη Συρία έχουμε μπλεχτεί ανάμεσα σε δύο πολιτικές διαδικασίες. Από τη μία έχουμε τη διαδικασία της Γενέβης, τις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο τη συνταγματική αλλαγή, τις ε, εκλογές ε, και την αποχώρηση από το καθεστώς του Ασάντ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σας το εξηγήσω αυτό πώς εξελίσσεται, αλλά υπάρχουν και, τις, υπάρχουν και οι συζητήσεις της Αστάνα που η Τουρκία, η Ρωσία και το Ιράν υποστηρίζουν που πηγαίνουν κάποιες φορές παράλληλα. Αυτές οι δύο διαδικασίες συνεχίζονται και προσπαθούν να φέρουν τους εμπλεκόμενους στο ίδιο τραπέζι για να βρεθεί μία ε, λύση βιώσιμη και διακανονισμός ε, ώστε να λήξει ο πόλεμος. Τώρα, ε, για τη διπλωματική και τη στρατιωτική πλευρά αυτής της σύραξης, δύσκολα μπορούμε να πούμε κάτι για το μέλλον. Αυτό που θα πρέπει όμως να πούμε είναι τι θα γίνει όταν τελειώσει αυτό. Πώς εμείς θα μπούμε στο ε, παιχνίδι. Αν δούμε τις προηγούμενες εμπειρίες μας, είναι σαν μια σκηνή από την ταινία Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον. Εδώ μιλάω για το Ιράκ στην ε, δεκαετία του 90, όταν είχαμε το Σαντάμ Χουσέιν στην Βαγδάτη, είχαμε την αυτόνομη κουρδική, κουρδική περιοχή στα βόρεια του Ιράκ και την περιοχή των Σιητών στο Νότο που εκπροσωπούσε την πλειοψηφία εντό της χώρας. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν έχουμε μια επανάληψη του ίδιου ε, σκηνικού και ίσως αυτό θα μας βοηθήσει να δούμε πώς θα είναι μετά η Συρία όταν θα είναι κατακαιρματισμένη και έτσι αποδιοργανωμένη. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας και κάποιες διαφορές. Στην περίπτωση της Συρίας, ε, το καθεστώς Ασάντ είναι πολύ πιο αδύναμο στρατιωτικά από ότι το καθεστώς Χουσέιν, τουλάχιστον προς το τέλος και ε, υπάρχει μεγάλη αύξηση της επιρροής εντός της Συρίας, κάτι που δεν συνέβη στην, στην περίπτωση του Ιράκ, παρά μόνο το 2003. Για την πολιτική, να πω τώρα, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτικών, πολιτιών, ε, ότι εμείς ε, δεν θέλουμε ρόλο στον Ασάντ ε, να μην υπάρχει στην κυβέρνηση. Θέλουμε ενωμένη Συρία. Αυτά είπε και ο Τίλερσον στη Γενέβη την περασμένη εβδομάδα όταν συναντήθηκε με τον Στέφαν Τεμιστούρα, τον ε, ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία. Όμως, ε, αν πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, ο στόχος για τη Συρία θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη λύση ε, και ένας διακανονισμός για τη λήξη του πολέμου, να υπάρχει μια σωστή ισορροπία ώστε οι γειτονικέ χώρες ε, να σταματήσουν να αλληλοσκοτώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία δεν θα χρησιμοποιούνται τακτικά τα χημικά και άλλα όπλα για να διατηρηθεί η ειρήνη και ε, το κερασάκι στην τούρτα και το καλό δηλαδή της υπόθεσης θα είναι ε, να επιστρέψουν και οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Δεν χρειάζεται καν να σας εξηγήσω εδώ γιατί. Επίσης, ε, να, αυτή, αυτός ο αποκλεισμός, η απομόνωση του καθεστώτος Ασάντ πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της δυτικής ε, πολιτικής. Πρέπει να έχουμε ευθυγραμμινισμένες κυρώσεις εμείς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα χημικά όπλα και τη χρήση τους. Ε, ειδικά για το περιστατικό Χανσεχίτε που είχαμε στις αρχές του έτους και ξεκίνησε τις αεροπορικές επιδρομές ε, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει εντός της Συρίας να υπάρξει μια ε, μετάβαση στη μελλοντική κατάσταση που δεν θα έχει επιστροφή. Θα πρέπει ε, εκεί που δρούν οι δυτικές ε, δυνάμεις, εκεί ακόμα που υπάρχει και η συμμαχία, όπου υπάρχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι παρακυβερνητικές οργανώσεις, οι δυτικές χώρες έχουν και θα πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο. Πρέπει να έχουμε τον ε, ίδιο κανόνα. Όλοι πρέπει να παίξουν ένα ρόλο μετά τον πόλεμο, αλλά το πώς αυτό θα ε, μοχλεύσει την διαδικασία είναι άλλο θέμα. Το να μην δίνουμε πόρους για την ανοικοδόμηση της Συρίας ε, στον Ασάντ και του συμμάχους του ε, είναι δυνατόν να συμβεί μεν, αλλά ε, και αν γίνει αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον ψήφισμα 254 των ε, Εθνών ε, σχετικά με τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να αφήσουμε όλη τη διαδικασία να εξελιχθεί για να δούμε ακριβώς πώς θα εφαρμόσουμε όλο αυτό το ψήφισμα. Επίσης, ε, από, τη σειρά, από την πλευρά σας θα πρέπει να πιέζετε τις κυβερνήσεις σας, να δείτε τι ακριβώς θέλουμε να δούμε στη Συρία, τι μας βολεύει, τι μας εξυπηρετεί και πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μια λύση η οποία θα βοηθά τους ανθρώπους στη Συρία κατά κύριο λόγο. Ευχαριστώ Άντριο Τίπλερ, για αυτή την ενημέρωση όσον αφορά την παρούσα κατάσταση στη Συρία. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν σχόλια, έχουν ερωτήσεις. ΕΛΚ, ο κ. Στετίνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας και τα αγγλικά βρίσκονται στο κανάλι 2. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά δεν αναφερθήκατε σε ένα θέμα που είναι σημαντικό και το ανέφερε ο πρόεδρος. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η ήττα στη Ράκα, αυτή η νίκη στη Ράκα κατά το ΆΕΣΙΣ. Πήγαμε στη Συρία και ξέρουμε πόσο οι Κούρδοι πολέμησαν στο Κομπάνε, έδωσαν μάχες. Και έχω την εξής ερώτηση. Ποιο είναι το μερτικό των Κούρδων, πόσο συνέβαλαν σε αυτή την ήττα στην Ράκα, στην περίπλοκη κατάσταση, ποια είναι η απόψη σας όσον αφορά το πολιτικό και διπλωματικό πεδίο, όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι προτιμάτε, να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις και σχόλια και μετά απαντάτε. Ωραία. Ο κ. Μποστινάρου για το σοσιαλιστικό, σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω αρκετές ερωτήσεις. Θα συγκρατηθώ και θα υποβάλω μόνο δύο. Πρώτη. Πόσο εφικτή είναι η νευτική διαδικασία στη Συρία. Πώς μπορεί να συμφιλιώσει τα δυσκόλως συμφιλιούμενα θέματα. Υπάρχουν πολλές πλευρές ε, με διαφορετικούς υποστηρικτές που συγκρούνται. Είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι θα επικρατήσει ειρήνη. Δεύτερον, τι ρόλο θα παίξει η Ρωσία στη Συρία. Γνωρίζοντας ότι η επιτόπια παρουσία τους ε, δεν αφορά μόνο τη Συρία αλλά και τη Μέση Ανατολή. Και έχει ανησυχητικές συνέπειες αυτή η παρουσία περισσότερες από αυτές που βλέπουμε και διαπιστώνουμε στη Συρία. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε στο μέλλον στη Συρία πώς θα αποφύγουν άλλη αποτυχία. Διότι εμείς σαν Ευρωπαίοι απουσιάζαμε. Απλώς κάναμε δηλώσεις παθιασμένες για την επιδείνωση της καταστάσεως, αλλά δεν κάναμε τίποτα να αποφύγουμε στην πράξη την επιδείνωση της καταστάσεως. Ευχαριστώ κύριε Μποστενάρο, του ECR. Ο κ. Μπέλτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μιλάει λίγο μακριά από το μικρόφωνο ο κ. Μπέλτερ και δεν τον ακούμε. Έχετε μια πολύ καλή ιστοσελίδα. Ο πρόεδρος επισημαίνει στον ομιλητή να μιλήσει κοντά στο μικρόφωνο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, έλεγα. Κύριε Τέιμπλερ, ε, το Ινστιτούτο σας το βρίσκω πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον και τα όσα γράφετε εσείς στην ιστοσελίδα για τη Συρία. Ο ρόλος της Τουρκίας με απασχολεί. Είναι ε, πραγματικά περίεργος. Γιατί δραστηριοποιείται σε μια περιοχή που είναι παρούσα και η Αλκάιντα με τα χρήρα Αλχάμ. Και τι κάνουν αυτοί, συνεργάζονται τώρα οι Τούρκοι με την Αλκάιντα. Είναι περίεργο, δεν σας φαίνεται σας. Υπάρχουν κινήματα που πρόσκυνται στην Αλκάιντα και συνεργάζονται με την Τουρκία. Υπάρχει μήπως κανένας δάκτυλος ε, του Κρεμλίνου για να βυθιστεί όλο και πιο βαθιά σε αυτό το βάλτο η Τουρκία. Και τι γίνεται με τους Κούρδους. υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμούς. Να εκχωρήσει η Δαμασκός, ας πούμε, το κεντρικό καθεστώς κάποιο είδος αυτονομίας στους Κούρδους της Συρίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται στο Κερκούκ τώρα οι Κούρδοι αλλάζουν συμμαχίες, εγκαταλείπουν ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε και στρέφονται προς τη Ρωσία. Επίσης υπολογίζεται η βοήθεια που χρειάζεται ε, για τη Ρωσία στα 150 δισεκατομμύρια. Και ορισμένοι τρίβουν ήδη τα χέρια τους για το πώς θα πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της χώρας. Και πώς επηρεάζουν τα πράγματα το Ιράν και η Ρωσία. Είμαι πολύ επιφυλακτικός για το μέλλον και την κατάσταση στη Συρία και ιδιαίτερα για το ρόλο της Δύσης Ευχαριστώ. Και τώρα για τους πράσινους. Λοχπίλα, συνάδελφε Πίλερ. Ευχαριστώ. στα αγγλικά. Ευχαριστώ και σας κύριε Τέιμπλερ. Ε, μιλήσατε για τη χρήση χημικών όπλων. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν τόσα πολλά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εκεί και εγκλήματα πολέμου. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Ε, είναι εγκλήματα που έχουν ε, διαπράξει και οι Ισλαμιστές, οι διάφοροι Ισλαμιστές, αλλά και το ίδιο το καθεστώς του Άσαντ στη χώρα μου, τη Γερμανία, νομίζω ότι έχουμε τώρα δύο ε, περιπτώσεις δραστών που ενδεχομένως να προσαχθούν ε, σε ένα διεθνές δικαστήριο. Αλλά δεν φτάνει αυτό από μόνο του. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, διστάζει να τους παραπέμψει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εσείς τι πιστεύετε τώρα στη μετάβαση ή μετά τη μετάβαση, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα πολέμου με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Άλλοι δύο μιλητές, ο κύριος Καστάλντο και μετά ο κύριος αφουζέρ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το διακεκριμένο αναλυτή για την παρέμβασή του. Έχω μια-δύο ερωτήσει. Διάβασα το άρθρο σας κύριε Τάμπλερ της 22 Σεπτεμβρίου του 2017 στο blog 8date, και αναφερθήκατε στην, ότι αναφερθήκατε στον Εφράτη και τη διέλευση των Συριακών στατευμάτων που ε, πέρασαν στην άλλη πλευρά του Εφράτη και ότι αυτό έχει συνέπειες. Και αυτή η διέλευση σήμαινε ότι έχουν κάτι υπόψη τους υπεύθυνοι στη Μόσχα στη Τεχεράνη και ίσως υπάρξει αντιπαράθεση με Ιράν, Ασάντ και Ρωσία είπα εναντίον αυτών. Ο Ασάντ με την υποστήριξη της Ρωσίας κατέκτησε περίπου 70% της επικράτειας. Νίκησαν όχι μόνο την ISIS και τους ζιχαντιστές κατά του καθεστώτος που υποστηριζόταν τη Σαουδική Αραβία από το Ριάντ. Τώρα τι περιμένετε από πλευρά ΣΥΠΑ. στρατηγική, διπλωματία. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, παρετήθηκε ο Λιβανός, Λιβανέζος Πρωθυπουργός κ. Χαρίρη ξαφνικά. Και ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλάν, ο πρίγκιπας, ανέρχεται στην ε, κυβέρνηση, κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό θα επηρεάσει την κατάσταση Συρία και την όλη υποστήριξη που δέχονται οι διάφορες ε, ομάδες που στήριζονται από τη ΣΥΠΑ και από άλλους. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο και ο Σαφχάουζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ διάφορα πράγματα μου έρχονται στο μυαλό και περιμένω την απάντησή σας. Πρώτον, ε, η αρχή της κυριαρχίας και των Ηνωμένων Εθνών. Η ανάμιξη, όταν δεν καλύπτεται από τα Ηνωμένα Έθνη, αποσταθεροποιεί και αποδυναμώνει την ίδια τη Δύση, εμάς τους ίδιους. Εδώ έχω υπόψη μου τις επεμβάσεις στο Ιράκ, στη Λιβύη αλλά και τη Συρία. Διότι εάν επεμβαίνουμε και προσπαθούμε να αναμειχθούμε με οποιασδήποτε αρχές ανθρώπινα δικαιώματα ε, που συχνά κρύβει ε, τον προσανατολισμό της εξουσίας και της ισχύω, δύσκολα μπορούμε να επικρίνουμε κάποιους άλλους που πράττουν τα ίδια. Η χώρα μου, ας πούμε, υποστήριξε την Αλ-Νούσρα και σήμερα μαθαίνουμε ότι ήταν τρομοκράτες αυτοί, τρομοκρατικές ε, οργανώσεις. Κάποιες αμερικανικές μαρτυρίες μας λένε τα ίδια ότι έμεσα η αμερικανική πολιτική ε, μάλλον υποστήριξε Ισλαμιστές. Κατανοώ ότι πίσω από αυτό υπήρχε η ιδέα αποσταθεροποίησης του Άσαντ. Αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, άραγε. Δεύτερον, από εκεί και πέρα μπορούμε πραγματικά να επικρίνουμε το Ιράν ή την Τουρκία, η οποία η ίδια χειραγωγεί τη χώρα με βάση τα δικά της περιφερειακά συμφέροντα ή τη Ρωσία. Θα πρέπει να ξαναβρούμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, αλλιώς δεν πρόκειται να κατευθυνθούμε προς μία λύση ειρηνευτική. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Δεν πρόκειται να έχετε πολιτική εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε μπορείτε να την επικαλείστε αν αγνοείτε την κυριαρχία του λαού αν θα πρέπει να φύγει ο Άσαντ να πέσει. Αυτό είναι ιστορικό πρόβλημα της Συρίας, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Οπότε, ας αφήσουμε εκεί τις διαδικασίες να ε, εξελιχθούν. Φανταστείτε τον κόσμο αύριο με μια Κίνα, μια Ινδία και άλλες δυνάμεις, όπου να θέλει κάθε μια να χειραγωγεί ένα μέρος του κόσμου. Πού βαδίζουμε, σε ποιο κόσμο πηγαίνουμε. Σας ερωτώ λοιπόν, δανειζόμενο στην περίπτωση της Συρίας, για σας ποιες είναι οι λύσεις της ειρήνης. Και τελειώνω με μια άποψη. Και εδώ μιλώ προσωπικά και όχι εκ μέρους της ομάδας μου. Εγώ τους συμπαθώ τους Κούρδους γενικά. Ιδού λοιπόν ένας λαός ο οποίος αγωνίστηκε, πολέμησε κατά της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας και είναι και ντόπιο δεν έχει έρθει απ' έξω, μπορεί να τον υποστηρίζουν απ' έξω, αλλά είναι λαός της περιοχής που υπάρχει εκεί. Και θα ήθελα την άποψή σας για την στήριξη στους Κούρδους ή τη μη στήριξη. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεφχάουζερ. Άλλα σχόλια? Όχι πολλές ε, πολιτικές απόψεις, ε, βρει φάσμα στην Επιτροπή μας. Ήρθε η ώρα να απαντήσετε σε όσο περισσότερες ερωτήσεις και σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις, καλύτε... τις γνώσεις που έχω αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά στο ρόλο των Κούρδων, στην πτώση της Ράκα να πω ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επανακατάληψη της πόλης από το Ισλαμικό κράτος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η επανακατάληψη της Ράκα από την SDF, της Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Ε, κάτω από την ίδια μπρέλα είχαμε και τους Κούρδους, YPG, και τις Άραβες που μάχονται σε αυτή την περιοχή, στην ίδια συμμαχία. Και μαζί κάτι που δεν περιμέναμε, ε, συνεργαστήκαν πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ε, συνεργασίας, ε, εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, αυτές οι δύο δυνάμεις βγήκαν στο προσκήνιο για να υποστηρίξουν τις δημοκρατικές δυνάμεις ώστε να επανακαταλάβουν τη ράκα και αυτό είναι στην ουσία ένα μοσαϊκό δυνάμεων ότι έχει απομείνει από τις δυνάμεις του Ασάντ. Αυτό είναι καλά νέα, όπως είπα. Βέβαια, στο μέλλον το πρόβλημα θα είναι η διατήρηση της πολιτικής πειθαρχία και αυτής ε, της ομπρέλας θα λέγαμε. Γιατί από τη στιγμή που ιτήθηκε ο Άισις και αν ιτηθεί και πλήρως, ε, οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ αυτών των ομάδων θα ανακατανεμηθούν. Δεν ξέρω αν θα, θα βιώσει, επιβιώσει αυτή η διαμόρφωση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, στην ουσία υποστηρίζουν τη σταθεροποίηση της περιοχής, ε, τις ε, συγκεκριμένες τοπικές δυνάμεις και τοπικές εκλογές. Αυτό θα βοηθήσει κατά τη γνώμη μας. Τώρα για το πόσο εύκολη είναι η πολιτική διαδικασία και πόσο εφικτή εξαρτάται από την πολιτική διαδικασία για την οποία μιλάμε. Κατά την γνώμη μου λοιπόν, πριν από 17 χρόνια στη Συρία και πολύ περισσότερο πριν στη Μέση Ανατολή, οι άνθρωποι ήταν λίγο πολύ οι ίδιοι. Ε, έτσι και οι κυβερνήσεις ε, δεν άλλαζαν ποτέ παρά μόνο αν έπρεπε, αν ήταν αναγκασμένοι. Αν ε, μπούμε λοιπόν σε διαπραγματεύσεις, δεν ξέρω ποια θα είναι η ανάγκη που θα κάνει την κυβέρνηση του ΣΑΝ να αλλάξει τις πολιτικές του και το ίδιο ισχύει και για την αντιπολίτευση, ειδικά αν έχουν ε, μαξιμαλιστικά αποτελέσματα πολιτικά. Ε, αυτή είναι η κατάσταση και αυτά συζητήσαμε και με τον Στέφαν Ντεμιστούρα. Ε, αυτά είναι που βλέπει παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνουν. Η διεθνής πίεση βέβαια λειτουργεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπουν ε, στο ίδιο στρατόπεδο και μαζί πιέσουν, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάτι. Αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι πιστεύαμε. Ο ρόλος της Ρωσίας σε αυτή τη διαδικασία, ξέρετε, δεν μπορώ πραγματικά να τον προβλέψω. Δεν ήθελα να μιλήσω εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά μπορώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και, τους, και τον περίγυρό του. Ε, είναι κάποια πράγματα που συζητούμε μαζί τους ε, και βλέπουμε ότι συμφωνούμε και εντάξει, ε, τους συμπαθούμε και θέλουμε και τους καλέσουμε και για μπάρμπεκιου. Από την άλλη πλευρά ε, δεν ισχύει το ίδιο. Αυτά συμβαίνουν. Ε, οι απόψεις των Ρώσων δεν είναι μονολυθικές. Θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, η έκβαση που περιμένουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πιέζουν είναι να έχουν μια στρατιωτική νίκη την οποία τελικά θα παρουσιάσουν και ως διπλωματική. Επίσης, ε, ε, φαίνεται ότι κάποιοι λένε ότι ίσως σιγά σιγά να θέλουν να μειώσουν την, παρουσίαση του, την παρουσία τους και την υποστήριξή τους εν ώψη των εκλογών ε, του χρόνου την Άνοιξη. Τώρα για το πώς οι Ευρώπη και οι Πολιτείες μπορούν να προβλέψουν και να προλάβουν μια νέα καταστροφή παρά τις θεωρίες και όλα τα άλλα που λέμε. Απλώς την ιστορία θα πρέπει να δούμε η πολιτική του Ομπάμα στη Συρία ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Δεν το λέω ε, γιατί έχω κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές ε, πεπιθήσεις, αλλά η αιμορρογία ανθρώπων, ο εξτρεμισμός, ε, ο σεχταρισμός, όλα αυτά είναι στοιχεία που βλέπουμε στην Μέση Ανατολή και δεν επηρεάζουν μόνο την περιφέρεια, αλλά την ευρωπαϊκή ασφάλεια γενικότερα η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ασφάλεια του κόσμου λοιπόν τα περιλαμβάνει όλα αυτά σχετικά με το ρόλο της Τουρκίας στο Ιντλίπ. Αν μαντεύω σωστά, αναφέρεστε σε κάποια βίντεο που, οι τουρκικές, που δείχνουν ότι οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις ε, προχωρούν και πηγαίνουν ε, και ε, ως συνοδεία στο STS. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες για να προχωρήσουν προς κάποιες ε, περιφέρειες και να παίξουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω ε, ε, εάν η Τουρκία υποστηρίζει το HTS και είναι θέμα πολιτικής τους, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι με την πάροδο του χρόνου ο στόχος του να ρίξουμε τον Άσαντ ε, κατέβηκε πιο χαμηλά στην ημερήσια διάταξη, δεν έφυγε, αλλά το Κρεμλίνο στην ουσία όθησε την Τουρκία σε αυτή τη σύραξη, πρώτον για να μπλοκάρει τις συριακές δημοκρατικές ε, δυνάμεις και το YPG συγκεκριμένα που θεωρούν εχθρό και δεύτερον για να μαχηθεί κατά του εξτρεμισμού εντός της Τουρκίας και να υπάρξει ε, μια, ένας πολιτικός διακανονισμός υπό του όρους που θέτει η Μόσχα. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον, ε, πολλά λέγονται. Εγώ νομίζω ότι αυτά που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όλοι κοιτάνε τη Συρία και βλέπουν τους ορούς από συντρίμια, τους εκτοπισμένους και όλοι θέλουν να πάνε για να κάνουν την ανοικοδόμηση της χώρας. Η Κίνα ε, μπαίνει στην ε, ουρά, το Ιράν, ε, όλες οι γειτονικέ χώρες, αλλά κανείς δεν θέλει να πληρώσει κάτι τέτοιο. Ούτε καν οι Ηνωμένε Πολιτείες, σας διαβεβαιώ, δεν θέλουν να να ανοικοδομήσουν, να πληρώσουν την ανοικοδόμηση μιας χώρας που κατέστρεψε ο Ασάντ, το Ιράν και η Ρωσία η δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ δεν είναι και η βέλτιστη, οπότε δεν πρόκειται να επενδύσουν σε κάτι, ε, εκτός αν υπάρχει μια καλόπιστη, ένα καλόπιστο πολιτικό αντάλλαγμα. Νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι ε, στο ίδιο μήκο κύματο κινούνται. Ε, δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν θα φέρει τίποτα η πολιτική διαδικασία, αλλά εδώ είμαστε τώρα. Τώρα για τα εγκλήματα πολέμου. Εξαιρετικό ερώτημα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν τέθηκε πιο νωρίς και πιο ξεκάθαρα αυτό το θέμα, πιο ευθέως. Ε, πολλοί θεωρούσαν ότι αν θέσουμε το θέμα των εγκλημάτων πολέμου πολύ νωρίς, ε, θα έχουμε λιγότερες επιλογές ε, για να κάνουμε τον ε, Ασάντε και τον άμεσο περίγερό του να φύγουν από τη χώρα. Για να πείσεις κάποιον να φύγει από τη χώρα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτή την απειλή. Καθώς όμως συνεχίζεται ο πόλεμος και οι φρικαλαιότητες και αυξάνονται οι απώλειες σε άμαχο πληθυσμό, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να δούμε το θέμα των εγκλημάτων πολέμου και να ανοίξουμε ζήτημα τέτοιο για τον πόλεμο στη Συρία. Υπάρχουν τόσοι πολλοί διεθνείς εταίροι που επεμβαίνουν εντός της Συρίας από διάφορα υπόβαθρα που μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί σε πολλές χώρες ε, για το πώς δηλαδή συμπεριφέρθηκαν. Άρα το να βρούμε έναν πολιτικό διακανονισμό στο τέλος θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Εγώ θα έλεγα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεμονωμένων χωρών να προχωρήσετε μεμονωμένα αυτή την προσπάθεια για τη λογοδοσία για αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Ε, υπάρχουν πολλοί στο καθεστώς του Ασάτ που θεωρούν ότι τα πράγματα θα επανέλθουν στην παρελθούσα κατάσταση. Αν στείλουμε το μήνυμα των εγκλημάτων πολέμου θα θέσουμε ένα όριο και θα καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό και ίσως να ξεκινήσει καλύτερα και να προχωρήσει καλύτερα η πολιτική διαδικασία. Γι' αυτό όλο αυτό το αφήνω στους, ε, νομικά, τους ε, δήμονες στα νομικά. Τώρα, τι να περιμένουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες και ειδικότερα τι διακυβεύεται μεταξύ Ασάντ Ιράν, Ρωσικής αεροπορίας κτλ. Ε, αυτό είναι λίγο ενδιαφέρον θα έλεγα, λίγο πιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι δυνάμεις υπέρ του Ασάντ, οι δυνάμεις του Ασάντ οι οποίες ε, επανακαταλαμβάνουν εδάφη από το Ισλαμικό κράτος μεταξύ άλλων όπως φαίνεται στο χάρτη. Αν ξαναδεί κανείς όμως καλά το χάρτη θα φαίνεται ε, η εικόνα σαν ένα μοσαϊκό δυνάμεων οι οποίες ε, μάχονται κατά του ISIS. Έχουμε όχι μόνο το Ιράν, αλλά πολύ, πολλές ξένες δυνάμεις. Έχουμε τους μισθοφόρους, τους Ρώσους που πρόσφατα συνέλαβε το Ισλαμικό κράτος, ε, την Ρωσική αεροπορία. Όλα αυτά ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουν στο να διατηρηθεί η ειρήνη σε μια περιοχή της Συρίας που είναι κυρίως σουνητική. Είναι πολύ νωρί για να το δούμε. Θα δούμε πώ θα, συμπεριφερθεί και, ε, θα συμπεριφερθούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, η ένταση που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας και Ιράν και Συρίας νομίζω ότι τελικά ε, μετά τον βομβαρδισμό του Χάν Σενχιούν από τον Τραμπ στις αρχές του έτους Ε, έτσι ώστε ε, να προχωρήσουμε ε, υπήρξαν οι αεροπορικές επιθέσεις από τις Ηνωμένες σε αυτή την περιοχή και υπήρξε μεγαλύτερη ένταση και τελικά έκλεισαν, κατέ, κατέριψαν οι Ηνωμένες σε ένα τζετ συριακό, αυξήθηκε η ένταση και ε, οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ξαφνικά έγιναν πιο αποτελεσματικές. Και φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την συμφωνία στην Ανατολική Συρία που έγινε για το ποτάμι τον Εφράτη, για το ποτάμι Εφράτη. Ε, υπάρχει αυτή η αναλογία με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι ακριβώς ε, το ίδιο αλλά και εδώ ε, είχαμε τους Ιρανούς από την Δύση και η Ρωσία και το SDF από την άλλη πλευρά. Όταν η Ρωσία πέρασε από τον ποταμό έφερε τις δύο δυνάμεις αντιμέτωπες. Ε, και αυτός ήταν ε, ένας από τους τρόπους που ήμασταν επιτυχείς ε, στο πώς μειώνουμε τις εντάσεις. Γιατί δεν είναι μόνο το να είμαστε εμείς και η Ρωσία μαζί κατά της Συρίας. Είναι και άλλα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε, να βρούμε μια πιο συγκεκριμένη λύση. Επίσης για την παρέτηση του Προέδρου Χαράρη. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε. Ακόμα αναρωτιέμαι, αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός χώρος μεταξύ του πολιτικού κράτους και του Χεσμολάχ έχει γίνει πιο μικρός η απόσταση δηλαδή μεταξύ τους. Η απώλεια της κάλυψης ε, ότι είναι Σουνίτες Άραβες ε, στην ουσία αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε εντάσεις μεταξύ Ισραήλ, Χεσμολάχ και Ιράν γενικότερα όσον αφορά το κομμάτι του Λιβάνου και της Συρίας. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πόλεμος, είναι λίγο υπερβολικό να το λέμε αυτό, όμως ε, πολλά μηνύματα στέλνονται με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος ε, που εξελίσσεται ο πόλεμος στη Συρία και στο Λίβανο δεν είναι αποδεκτός από το Ισραήλ και φυσικά θα υπεραμενθούν των συμφερόντων τους. Τώρα για την ε, κυριαρχία των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει ένα ολόκληρο μείγμα τρόπων με τους οποίους ο καθένας δικαιολογεί την εμπλοκή του στον πόλεμο της Συρίας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, και αυτή ήταν απόφαση του Ομπά, αποφάσισαν να μην παρεμβούν στη Συρία λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως παρενέβησαν για να καταδιώξουν το Ισλαμικό κράτος σύμφωνα με την διακήρυξη ναι, του άρθρου 51 της Δημοκρατίας του Ιράκ. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, λοιπόν, ε, και πολλοί, οι Ηνωμένε Πολιτείε και πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή είστε στη Συρία γιατί ο Μπασάρα Λασάντ ε, έχασε τον έλεγχο και μια ε, γειτονική χώρα μας ζητά να μπούμε και να φέρουμε μια οργάνωση σε αυτά τα εδάφη. Η οργάνωση λοιπόν αυτή, αυτή τη στιγμή ε, συρρυκνώνεται και δεν υπάρχει και νομική υπόσταση και γι' αυτό το πώς θα το διατηρήσουμε είναι μεγάλο ερώτημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπως γνωρίζετε, δικαιολόγησαν τον πόλεμο στη Συρία ε, σύμφωνα με την νομοθεσία που έχει μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου και σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό. Υπάρχουν όμως πολλά, ε, πολλοί παράγοντες που παρεμβαίνουν τώρα στη Συρία και οι γειτονικέ χώρες και η Συρία δυστυχώ έχει γίνει ένα παιχνίδι χωρί σύνορα. Και υποπτεύομαι ότι είτε θα, έχουμε μια πιο καλή κυβέρνηση, πιο οικουμενική κυβέρνηση στη Συρία, είτε θα έχουμε μια κατακαιρματισμένη Συρία η οποία δεν θα έχει τη νομική ε, υπόσταση ώστε να προχωρήσει. Είναι ανοιχτό αυτό το σύντημα. Και το τελευταίο που θέλω να πω έχει να κάνει με το καθεστώς Ασάντ αν είναι εσωτερικό θέμα. Κοιτάξτε, αυτό θα είναι τελικά το αποτέλεσμα της πολιτικής διαδικασίας είτε στη Γενέβη που έχει να κάνει με την αλλαγή του συντάγματος, τις εκλογές κτλ. είτε όχι. Ε, όμως, όπως και να έχει, ε, όλοι καταλαβαίνουμε πως ε, η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών ευρωπαϊκών χωρών για την έκβαση αυτής της σύραξης βασίζεται στη συμπεριφορά μιας υπεύθυνης κυβέρνησης εντός της Συρίας ε, η οποία θα έχει σωστές σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες και θα διάγει μια καλή εσωτερική πολιτική. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε διαφορετικό δρόμο ως προς αυτό. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι η επιρροή των ΗΠΑ στη Συρία δεν ήταν ποτέ μεγάλη. Ποτέ δεν υπήρξε η Συριακή Αραβική Δημοκρατία σύμμαχος των ΗΠΑ, ούτε και θα γίνει πιστεύω. Όμως ε, η βασική, η πρωταρχική σημασία ε, της Συρίας είναι γεωγραφική. Είναι σαν ένα ε, σπιτάκι στο κέντρο μιας γειτονιάς που ό,τι και να του συμβεί επηρεάζει όλα τα γειτονικά σπίτια, όλη τη Μέση Ανατολή λοιπόν. Το να βελτιώσουμε λοιπόν τη λογοδοσία και δεν μιλάω για την δημοκρατία, είναι ένα αξιοθαύμαστο ιδανικό η δημοκρατία και την υποστηρίζω και εγώ όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλο τον κόσμο, αλλά χρειάζονται πολλά βήματα να γίνουν μέχρι να φτάσουμε σε αυτό. Ε, θέλουμε κάτι πιο αντιπροσωπευτικό και πιο ειρηνικό. Προς το παρόν δεν έχουμε ούτε καν αυτό. Έχουμε ενδιάμεσες λύσεις με ημίμετρα με πολύ λίγη πολιτική βούληση από οποιαδήποτε πλευρά να παρέμβει ε, το οποιοδήποτε, οποιοδήποτε στη Συρία. Και αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι η τάξη παρά η σταθερότητα. Αυτό είναι που έχουμε ε, στο μυαλό μας τώρα και γι' αυτό συζητάμε με τη Ρωσία. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω για τους Ρώσους, ε, θα μιλήσω για τους Αμερικανούς, για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Πρώτα έρχεται η σταθερότητα και μετά η τάξη. Όμως οι Ρώσοι το βλέπουν ανάποδα. Πρώτα η τάξη και μετά η σταθερότητα. Και μάλλον και οι δύο να κάνουμε λάθος. Ίσως κάνουμε λάθος, ίσως κάπου στη μέση να είναι η αλήθεια το να συνεργαστούμε προς ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο. Αν φτάσουμε όμως στην προηγούμενη κατάσταση, στην ουσία θα είναι σαν να ρίχνουμε λεφτά σε μια μαύρη τρύπα, σε, στις τσέπες ανθρώπων που δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Αν έχουμε όμως ένα σύστημα πιο σταθερό και ε, άξιο εμπιστοσύνη ε, θα λύσουμε πολλά προβλήματα για τις δυτικές χώρες και για τις ε, Ηνωμένες Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τέιμπλερ που απαντήσατε όλες τις ερωτήσεις, καλύψατε τις ερωτήσεις, τα θέματα που έθιξαν τα συγκεκριμένα μέλη της ΑΦΕΤ. Έχουμε κάνα δύο λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Ερώτηση λοιπόν. Υπάρχει κάποιος άλλος που ζητά το λόγο. Ο κ. Μποστινάρου πρώτος. Όχι, όχι, συγγνώμη. Τσάρλς Τάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια-δύο ερωτήσεις. Πριν από πέντε χρόνια, ίσως αφελώς, ζήτησα να αποκλειστεί ο εναέριος χώρος κάποιες περιοχής. Μου είπαν ότι ήταν στατιωτικά ανέφικτο τότε. λόγω του συστήματος του αντιπυραυλικού του Άσαντ και των διαφόρων συστημάτων που είχε και ότι κανείς δεν θα είχε τη δύναμη της Ειρητική να το εφαρμόσει. Μπορούσε να γίνει τώρα, με την πάροδο των ετών, να το δούμε αυτό. Θα είχαν σωθεί εκατοντάδες χιλιάδες ε, άνθρωποι εάν μπορέσαμε να τον ρίξουμε τώρα πριν μπουν στο παιχνίδι όλοι οι τζιχαντιστές του κόσμου. Άλλη ερώτηση. Οι Κούρδοι. Είμαι πρόεδρος ε, της ομάδας ε, που ασχολείται με το θέμα του Κουρδιστάν. Έγινε το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία. Εκεί οι Σιήτες, η κυβέρνηση της Βαγδάτες και οι Ιρανικές δυνάμεις κινήθηκαν προς το Κυρκούκ. Αν νικηθεί επιτόπου το ISIS, ο Άσαντ θα στραφεί κατά το STF και του YPG, των φυσικών συμμάχων των Αμερικανών, υπό τουρκική πίεση που είναι και μέρο του ΝΑΤΟ. Αν γίνουν αυτά, ποιο είναι το μέλο των Κούρδων στη Συρία και στο γειτονικό Ιράκ. Ποιο θα του αναγνωρίσει το δικαίωμα να έχουν τη δική του χώρα. Μπορεί να πιεστεί ο Ασάντ, ούτω ώστε να δημιουργηθεί μια ομοσπονδιακή Συρία που θα δώσει μεγαλύτερη αυτοδυναμία και δυνατότητα αυτοδιοίκησης στους ε, Κούρδους. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ο κ. Χόιντ είναι επόμενος. Ευχαριστώ. Είπατε κάτι πριν. Αφορούσε την πολιτική του Μπαράκ Ομπάμα στη Συρία. Δεν είπατε ότι ήταν καταστροφική μεν, αλλά το υπονοήσατε αναφερόσασταν στην ε, πολιτική της κόκκινης γραμμής και ίσως όχι μόνο σε αυτό. Παρακολουθούσα τότε στενά τις εξελίξεις. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει. Η πολιτική της χωριστικής, της κόκκινης γραμμής δεν οδήγησε πουθενά. Τι άλλο να κάνει όμως. Αυτή ήταν η μεγάλη ερώτηση τότε, η σημαντική ερώτηση. Είχαν κουραστεί και οι Αμερικανοί, δεν ήθελαν να παρασυρθούν σε άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προσπαθώντας να ξεμπερδέψουν από το Αφγανιστάν. Ποια είναι η άποψή σας, τι θα προτείνατε τότε. Και δεν ξέρω αν είχατε απόψεις που τις είχατε εκφράσει τότε. Ευχαριστώ κύριε Φράιντ. Άλλους? Δεν έχουμε άλλον. Ο κύριος Τέιμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι σαν να κοιτάμε στο παρελθόν, σε κρυστάλλινη σφαίρα. Δεν ξέρω αν κοιτά προς το μέλλον ή το παρελθόν σε κρυστάλλινη σφαίρα. Κάνουμε υποθέσεις για την ζώνη απαγόρευσης των υπερπτήσεων. Κάποτε, ε, δεν ξέρω αν ήταν εφικτό, θα έσωσε ζωές μια απαγόρευση υπερπτήσεων η Συριακή αεροπορία έπλητε στόχους πριν παρεμβούν οι Ρώσοι. Ε, βομβάρδιζε την αντιπολίτευση, νοσοκομεία, φούρνους βομβάρδισε. Έτσι θα προστατευόταν κάποιοι. Θα υπήρχε κάλυψη. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Δύο προβλήματα υπήρχαν για μια τέτοια παρέμβαση. Το πρώτο πρόβλημα. Το πολιτικό περιβάλλον στις περιοχές αντιπολίτευσης η αντιπολίτευση ήταν πιο κατακαιρματισμένη τότε. Δεν εκπλήσει αυτό. Υπήρχαν διχασμοί. Ε, επλήττοντο στα δυτικά αυτές οι περιοχέ. Αλλά η επαγόρευση υπερπτήσεων σε κάποιε περιοχέ τη Συρίας θα παρήχε κάποιο βαθμού ανθρωπιστική προστασία. Θα υπήρχε μια βάση για πολιτική διαδικασία σε αυτές τις περιοχές. Εγώ ήμουν διστακτικός εγώ δεν πιστεύω ότι θα λύναμε όλο το πρόβλημα της Συρίας και του πολέμου. Μάθαμε το Ιράκ ότι η επίλυση προβλημάτων άλλης χώρας είναι πολύ δύσκολο. Κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπήρχε κάποια δυνατότητα σε κάποιες περιοχές. Θα λειτουργούσε τελικά. Πώς θα επηρεαζόταν ο πόλεμος, δύσκολο να πει κανείς. Δεν γνωρίζω. Δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος. Τι ξέρουμε όμως ότι ακολουθεί θύσα πολιτική, και εδώ αναφέρομαι στην Ουάσιγκτον, ε, και τι πολιτικές του Πρόεδρου Ομπάμα, οι πολιτικές αυτές οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση. Οι ΙΠΑ έχουν ευθύνε για τις εξελίξεις. Και όχι μόνο για τα ανθρωπιστικά προβλήματα, αλλά και για το πώς ξέσπασε και επεκτάθηκε και ο Άισις και η Αλκάιντα. Υπήρχαν οι τάσεις από την αρχή της εξέγερσης σε όλες τις περιοχές της Συρίας. Εδώ μιλώ ως Αμερικανός. Οι τρομοκρατικές υποθέσεις που εντοπίστηκαν από τη ΣΥΠΑ αυξανόταν και γεγαντωνόταν σε κάθε περιοχή από την αρχή της σύραξη. Στην πράγμα του χρόνου αυξήθηκε η δύναμή του. Δημιουργήθηκε μια μαύρη τρύπα. Ε, πόλεμος για αντιπροσώπων, ε, συγκρούσεις ομάδων ε, και όλα αυτά οδήγησαν στην καταστροφή όσον αφορά το Συριακό λαό. Και τελικά αποδυναμώθηκε αποδυναμώθηκαν και οι σχέσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο ρόλος των Κούρδων, ένα από τα μεγάλα προβλήματα στα οποία βασίστηκαν και επικρίσεις που ακούστηκαν για την πολιτική των ΗΠΑ, ποιο ήταν, ότι ΙΠΑ στήριξαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Για πολλούς λόγους έγινε αυτό. Η ΗΠΑ είναι σε συμμαχία με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και είναι παραδοσιακό σύμμαχο των ΗΠΑ και θεωρεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις σαν κάλυμα για το ΠΚΚ που θεωρούν ε, ότι είναι ε, αντίπαλος. Η Αμερική υποστήριξε το SDF αντίθετα στις επιθυμίες της Τουρκίας. Αλλά υπήρχε ανησυχία ότι η συνεχή στήριξη των Κούρδων από πλευρά ΣΥΠΑ θα ήταν εις βάρος των θέσεων της ε, Τουρκίας που θα έχανε και έναντι της Ρωσίας. Νομίζω ότι είπα θα εξακολουθούν να υποστηρίζουν το SDF για σταθεροποίηση. Πολιτικές στοιχείες. Εδώ είναι περίπλοκα τα πράγματα. Έχουμε τον κουρδικό λαό στο σύνολό του που διαιρείται πολιτικός σε διάφορες ομάδες όπως ξέρετε. Το πιο δύσκολο πρόβλημα πολιτικό για τους Κούρδους είναι να συντονιστεί με τις ε, δυτικές προσεγγίσεις. Το πρόβλημα είναι με το YPG που έχει μια ιδεολογία που οδηγεί σε περιορισμό πολιτικής συνεργασίας. Χρησιμοποιούν, είπα, αυτή την οργάνωση για προσπάθεια που καταβάλλεται για την ήττα του ISIS και πολλοί στη Συρία το πιστεύουν, στηρίζουν για την ώρα τις περιοχές που ελέγχονται από το SDF. Τώρα να πιεστεί ο Άσαντ. Όπως και οποιοδήποτε άλλο στην περιοχή και ο Άσαντ χρησιμοποιεί ραβδί και καρότο, ένα μείγμα των πολιτικών αυτών. Ξέρω ότι αυτό είναι χιλιοϊπωμένο. Τι παρατηρούσα με την πολιτική στη Συρία. Και ίσως να αλλάξει αυτό βέβαια. Παρατηρούσα ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούμε μία το ξύλο και μία το καρότο. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε μόνο καρότα και μόνο ραβδιά και γι' αυτό ε, δεν καταλαβαίνει, δεν εκπληκτόμεθα που δεν πετύχαμε κάτι. Οι ΕΠΑ ε, θέλουν να πιέσουν μια διευθέτηση χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία της εργαλειοθήκης και όχι ε, ένα άλλο μείγμα. Θα δούμε. Περιγράφει και μια πολιτική για το Ιράν. Την περιγράψε ο πρόεδρο. Η πολιτική για τη Συρία αναμένεται. Σχετίζεται με την πολιτική για το Ιράν. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώ θα διαμορφωθεί. Οι, Ευρω... Οι να καταπολεμήσουν το ISIL. Η πολιτική θα λήξει, θα μπούμε σε νέα φάση. Και όταν μπούμε στη νέα φάση θα δούμε τι θα γίνει με το Ιράν και πώς θα επηρεάσει τη νέα στρατηγική θέση του Ιράν στη Συρία. Τώρα, η κόκκινη γραμμή του Προέδρου Ομπάμα. Σε κάποιες φάσεις του πολέμου, αρκετές από αυτές, οδηγηθήκαμε σε αυτή την καταστροφή πριν την κόκκινη γραμμή του Ομπάμα. Πήρε μια απόφαση το καλοκαίρι του 2012 να μην εξοπλιστεί η Συριακή Αντιπολίτευση, ο ελεύθερος Συριακός στρατός όπως απεκαλεί δεν αποφασίστηκε οι περιφερικοί σύμμαχοι να το κάνουν αυτό, να του εξοπλίσουν χωρί εμά. Άρα βγήκαν εκτό οι ΙΠΑ, μέχρι αργότερα. Επανήλθαν οι ΙΠΑ, ξαναμπήκαν στην αίθουσα. Και ξαφνικά χρήματα πήγαιναν παντού σε διάφορε ομάδε στην ε, Συρία που επιδίνωναν ε, τον διχασμό στη Συριακή αντιπολίτευση. Και κάποια από τα χρήματα έπεσαν στα χέρια ομάδων που θεωρούνται εξτραμιστικέ. Και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρώπη. Αυτή ήταν ατυχέστατη εξέλιξη έπρεπε να το αναμένουμε. Διότι η περιοχή βλέπει αυτή τη ομάδα διαφορετικά από ότι εμεί. Και άλλη απόφαση μετά ήρθε. Ταυτόχρονα μάλλον. Να καθοριστεί αυτή η κόκκινη γραμμή. Ιδιαίτερα κακή απόφαση. Τάχιστα, μετά τον καθορισμό της κόκκινης γραμμής, περίπου Αύγουστο του 2012 νομίζω, Ιούλιο-Αύγουστο κάπου εκεί, το καθεστώς Άσαντ άρχισε, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, και αποδείχθηκε μετά, ας χρησιμοποιεί χημικά όπλα με χαμηλή συγκέντρωση. Και το χρησιμοποιούσε όλο και πιο πολύ για να δει. Θα τον εντοπίσουμε, θα τον εντοπίσουμε, δοκίμαζε. Το Μάρτιο του 2013 λοιπόν, ο εκπρόσωπος της κυβερνήσης Ομπάμα είπε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή. Γιατί τώρα πρόεδρος αποφάσισε από το Μάρτιο του 2013 και τον Αύγουστο 2013 να μην προετοιμάσει το αμερικανικό κοινό για να επιβάλλει την κόκκινη γραμμή. Δεν ξέρω γιατί περίμενε. Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Κάποιες θεωρίες σχετίζονται με την τάση του να χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη, στρατιωτική ισχύ. Κάποιοι λένε ότι είπα είχαν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν και περιοριζόταν όσον αφορά τη στρατιωτική τους δράση στη Συρία εξ αυτού. Το να μην επιβληθεί κόκκινη γραμμή, εγώ ξέρω ότι έβγαλε εκτός της ΙΠΑ. Δεν μπορούσαν πλέον οι ΙΠΑ να επηρεάσουν τον πόλεμο. Και ε, αυτό έδειξε σε πολλούς από εσά και στους συμμάχους στη Μέση Ανατολή και στην Αποανατολή ότι δεν υπήρχε αμερικανική αποφασιστικότητα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις απορρέων της συνθήκες μας. Και αυτό είναι κατανοητό. Και τελικά κόστισε αυτό τη ΣΥΠΑ. Ένα κάτι είναι προσδόκητο αλλά και ενδιαφέρον επί Προέδρου Τρόμπ μόνο θα εφαρμοζόταν αυτή η κόκκινη γραμμή, αντιστρέφοντας πλήρως τα αναμενόμενα. Αυτά που περίμεναν θα είναι η πολιτική Τραμπ στη Συρία. Γιατί? Διότι όταν είσαι στη θέση του Προέδρου και βλέπει τα γεγονότα και τα πραγματικά στοιχεία, η χρήση του Σαρίν στη Συρία, αφού είχαν δεσμευτεί ε, με τους Ρώσους να καταστραφούν τα αποθέματα, εξόργησε αυτό τον Πρόεδρο. Και αυτό οδήγησε σε στρατιωτικό πλήγμα στη βάση του handshake. Επιβάλλεται η κόκκινη γραμμή. Τώρα, αν αυτό θα οδηγήσει στην λήξη της χρήσεως χημικών όπλων στη Συρία, δεν ξέρω. Οι ΙΠΑ δεν μπορούν να λύσουν τον πόλεμο Συρία, ούτε εσείς. Οι ΙΠΑ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του πολέμου όμως. Και δυστυχώς χάσαμε ε, πολλά κομβικά σημεία, ώστε να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άντρου Τέβλου που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, εξωτερικών υποθέσεων σήμερα το απόγευμα. Από πρώτο χέρι, πολύτιμα τα στοιχεία που μας δώσατε και καλή τύχη σε επόμενα καθήκοντά σας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουμε μια μικρή διακοπή μέχρι τις 5 και 4, ένα τέταρτο διάλειμμα και θα ακολουθήσουν ψηφοφορίες για τις εκθέσεις που έχουμε προβλέψει. Αντεβού στις 5 και 4.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 ήθελα να περάσουμε στις ψηφοφορίες μας, στο σημείο υπαριθμών 7. Θα θέλατε να καθίσετε κάποια στιγμή, παρακαλώ. Και όσοι δεν θέλετε να καθίσετε, παρακαλείστε να αποχωρήσετε. So we come to item number seven, the... Σημείο 7, λοιπόν, ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Ο εισηγητής δεν θέλει να πει τίποτα. Να ψηφίσουμε λοιπόν αμέσως. Ο κύριος Νάρτ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω μια προφορική τροπολογία στο σημείο 249 και θα ήθελα σύντομα να εξηγήσω ότι η κατάσταση στην Κολομβία δεν χρειάζεται απλώς στήριξη στην νευτική διαδικασία αυτή τη στιγμή, αλλά και έκκληση προς τις ΦΑΡΚ έτσι ώστε να δώσουν στα θύματα την περιουσία τους που έχουν αποκτήσει από λαθρεμπόριο ναρκωτικών και μπορούν να βοηθήσουν στην πάταξη του λαθρεμπορίου ε, δίνοντας προφορίες για τα δίκτυα στα οποία έχουν συμμετάσχει. Αφού είπαν ότι θέλουν να γυρίσουν σελίδα από αυτή τη μαύρη περίοδο της ιστορίας και να εμπλακούν στο πολιτικό παιχνίδι, στην κανονική διαδικασία, χωρίς ε, θησαυρού και χωρίς ε, ναρκοχρήματα. Και καταθέτω αυτή την προφορική τροπολογία για τη σταθεροποίηση στην περιοχή και ζητούμε, απαιτούμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία ε, των ΦΑΡΚ, μεταξύ αυτού και ο θησαυρό που έχουν αποκομίσει από το ε, λαθρεμπόριο, να ε, δοθούν στα θύματα της σύρεξης. Επίσης, να δώσουν πλήρη πληροφόρηση για τα εγκληματικά καρτέλ και τα δίκτυα. Αυτή είναι η προφορική μου τροπολογία για την Κολομβία, λοιπόν, και την παράγραφο 249. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος... Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, εγώ τρελαίνομαι για εκπλήξεις, αλλά ε, προσπαθώ τώρα να το χειριστώ όσο γίνεται καλύτερα αυτό που μου λέτε. Ορίστε. Well... Κάτι λέει ο κύριος Στανόκα, αλλά δυστυχώς δεν ακούγεται. Στο κύριο Νάρτ απευθύνομαι. Κοιτάξτε, ε, από την αρχική σας τροπολογία θα μπορούσα να υποστηρίξω τη φράση που λέει «Επαναλαμβάνει τη στήριξη της ενευτική διαδικασία στην Κολομβία που είναι αποφασιστική για το μέλλον των Κολομβιανών και τη σταθεροποίηση της περιοχής». Αυτό μπορώ να το εγκρίνω και να το υποστηρίξω. Όπως επίσης και το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ΦΑΡΚ συμπραγματευμένων του Δησαυρού από το λαθρεμπόριο ε, ναρκωτικών ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, προς όφελος των θυμάτων. Θα μπορούσα να το δεχτώ, αν και δεν μου αρέσει η διαδικασία, ο τρόπος που μου το θέτεται. Συμφωνείτε εσείς οι υπόλοιποι. Και σε ποιο συμβιβασμό θα μπει στο 13α. Ωραία. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, σοσιαλιστές και δημοκράτες. ECR, ε, φιλελεύθεροι φυσικά, συμφωνείτε. Καλώς. Προχωρούμε λοιπόν και ψηφίζουμε ευθύ αμέσω. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1. Ψηφί υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Όχι, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 35 ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος έτσι για να ζεσταθούμε προθέρμαση. Αρχίζει ψηφοφορία. Είναι. Εγκρίνεται. 28-8. Συμβιβαστική 3. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, όχι. Προηγουμένως έχουμε την τροπολογία 95 και σε δύο τμήματα μάλιστα. Τμήμα πρώτο, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ φωνές. Έλεγχο θέλετε, καλώς. Ε, ελέγχουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική υπαρθμόν 6 κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 113 Είπε. κατά αποχές αυτό θέλει επαλήθευση παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απέριφθη. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 7α και η προφορική τροπολογία παριθμό 1 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίθηκε. Ωραία. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ. Την 142 επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Όχι, υπάρχουν και άλλες τροπολογίες προηγουμένως που πρέπει να ψηφίσουμε. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. 222 της κυρίας Βάουτμανς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Καλά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 224. Της κυρίας Λόιζινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 227 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεκ. 2.27 λοιπόν, επαθεύουμε την απολογή αυτή, ψηφοφορία. Πέρασε. Wow, εγκρίθηκε. Συμβαστική 13 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε στην 242 της κυρίας Βάουτμαν. Ψήφιπε. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. 2.42 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα ερχόμαστε στη 13α, συμπεραμβαλωμένη τη προφορική τροπολογία του κυρίου Νάρτ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 264 του κύριο Μέζεριτς είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 266 καταπίπτει, οπότε θα πάμε στη 262 του κυρίου Πρέντα Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική όχι, διορθώνει πρόεδρος 36 ε, Λόζινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές. Παρακαλώ να την ελέγξουμε. Αρχίζει ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία υπαρίθμη 21. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές αναφορές, citations, 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Καλώς. Στη 2 λοιπόν, αιτιολογική αναφορά 2, αρχίζει ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Ένας. Ωραία. Πέρας. Απέριφθη. Προχωρούμε. Ε, τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει μια συμβαστική υπαριθμή 20 που εγκρίθηκε, οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ψηφίζουμε το σύνορο λοιπόν της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία παρακαλώ. Ένας συνάδελφος δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πάμε στο, στο σημείο. Παρακαλώ κυρία Λούζινγκ. Εξ ονόματος της ομάδας μας έχουμε συντάξει έκθεση μειοψηφίας και την έχουμε ήδη καταθέσει στη γραμματεία. Ευχαριστώ κυρία Λούζινγκ. μία 8 ετήσια έκθεση ετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και έρευνας. Μάιχαλ Γκάλερ είναι ο συγκητής. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε απευθείας. So we come to compromise. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική... Ε, τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 σε δύο τμήματα. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 37. Κυρία Λούζινγκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 39. Πίτσουλα υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 49. Cover υπέρ. Κατά απόχέ. απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αν εγκριθεί, πάμε στην προφορική τροπολογία παριθμών 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 και 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. 114 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 117 άρχεται η ψηφοφορία ο ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας απορρίπτονται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 καταπίπτει, 131 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 133 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 141 και 142, 140 142 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται, 143 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται.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 158 μέχρι 163 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 164 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 165 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 184 και 185 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 187 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 198 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 199 και 200 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 201 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για τη 203. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, α, εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206, 207 και 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 Ακρίμα που καταπίπτει 239, ήταν έξοχη τροπολογία. 240 υπέρ, κατά αποχές, α, 241 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 242 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 243 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 241 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 245 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 246 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 247 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 248 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 251 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 255 υπέρ, κατά αποχές Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 279. Πέιτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ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 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Και Λούζη. Um, uh, η ομάδα μου έχει γράψει μια έκθεση μειοψηφίας και την έχει στείλει ήδη στη Γραμματεία. Ευχαριστούμε την κυρία Λετζίνκ και πάμε τώρα στο σημείο 9. Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη. Πρώτα να δώσω τον ρόλο στον Αρνό Ντανζάν, τον εισηγητή μας, για να μιλήσει σχετικά με την ε, συμφωνία που έγινε ε, διοργανικά για το θέμα αυτό συμβιβασμός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω ότι οι δύο απαιτήσει που είχαμε όταν στον τριμηρέγη διάλογο κάναμε τη διαπραγμάτευση ικανοποιήθηκαν και οι δύο. Η θέση του Κοινοβουλίου λοιπόν αναγνωρίστηκε ειδικότερα με μια κοινή δήλωση η οποία θα επισυναφθεί στο κείμενο. Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο που έχει να κάνει με τη χρήση του εργαλείου συνεργασίας ε, και ανάπτυξης για την ε, χρηματοδότηση αυτής της ε, δράσης. Ικανοποιήθηκε λοιπόν το αίτημά μας το αρχικό και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ευχαριστώ την ομάδα για την εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ Αρνό. Να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που έχεις κάνει ως εισηγητής. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Είχαμε εξαιρετικές διαπραγματεύσεις, ειδικά με το Συμβούλιο. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι. Όχι, οπότε Άρχεται η ψηφοφορία. ...36 παρόντες πέρα της ψηφοφορίες και η 30 εγκρίνεται με 27 υπέρ και 7 κατά. Στις 29 και 30 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον ε, Δεκέμβρη-Γενάρη θα γίνει η δημοσίευση στην εφημερίδα την επίσημη. Ε, για τα διάφορα δεν υπάρχει κάτι. Στις 13 Νοεμβρίου στις 7.30 θα έχουμε την επόμενη συνάντησή μας στο Στρασβούργο. Πέρα στη συνεδρίαση, καλό βράδυ.